Uh, um, καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, φυσικά συνεχίζουμε τις ε, συνεδριάσεις των Επιτροπών. η σημερινή όμως είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί έχουμε κοντά μας τον Μιγκέλα Αρίας Κάνιέτε, Επίτροπο για την Κλιματική Δράση και την Ενέργεια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν μαζί του σήμερα το διαρθρωμένο μας διάλογο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Επίτροπος Κανιέτε προσεκλήθη ε, στην Επιτροπή Ήτρε, όχι για πρώτη φορά, και έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια, το χρονοδιάγραμμα, το συντονισμό και Βεβαίως, κύριε Επίτροπε, αν μπορούσατε να μας δώσετε και κάποιες προοπτικές για το πρόγραμμα εργασιών του 2018, θα σας ήμασταν ευγνώμονες. Γιατί θέλουμε και εμείς να προετοιμαστούμε για τις επόμενες προεδρίες, <coughs> μετά την Εσθονική δηλαδή, την Αυστριακή και ούτω καθεξής. If ε, μήπως θα είχατε την καλοσύνη να αναφερθείτε και στο νέο νομοθετικό σας πρόγραμμα. Αν έχετε βέβαια, αν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιο πρόγραμμα, γιατί ήδη έχουμε επιτάπητος 8 νομοθετικές προτάσεις ε, προς συζήτηση από την Ενεργειακή Ένωση και σημαντικό αριθμό προτάσεων και για την ε, ψηφιακή ένωση, ένωση ψηφιακής αγοράς. Αλλά είμαστε έτοιμοι και θα μπορούσαμε να εργαστούμε ακόμη πιο σκληρά. Επίσης, ε, έχουμε δρομολογήσει την εξέταση των 8 νομοθετικών προτάσεων με βάση το δικό μας φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με την κοινή διακήρυξη που προσυπογράψαμε στις αρχές του έτους. Κύριε Επίτροπε, έχουμε σχεδόν παραγνωριστεί θα έλεγα. Είμαστε τόσο εξοικειωμένοι που δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Να σας δώσω το λόγο απλώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριοι συντονιστές, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερος που ξανασυναντιόμαστε και σήμερα για το διαρθρωμένο μας διάλογο για να βοηθηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2018. Το 2017 μέχρι στιγμή, ήταν χρονιά εφαρμογής των προτάσεων που ε, εμπίπτουν στο πακέτο ασφάλειας του ανεφοδιασμού που υπευλήθη το Φεβρουάριο του 2016 και ακολουθεί τα πακέτα του περασμένου Νοεμβρίου. Και το πακέτο για την καθαρή ενέργεια είναι επίσης ε, ένα φιλόδοξο και μεγαλοεπίβολο πακέτο που ε, θα περιλάβει νομοθετικές προτάσεις για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις μας από τη Συμφωνία των Παρισίων. Ξεκινώντας με την με το σύστημα εμπορίας εκπομπών μετά το 2020, με τον επιμερισμό των ε, ε, προσπαθειών για τη μείωση εκπομπών στα κράτη-μέλη και το LULUCF. Επίσης, ε, το Φεβράριο του 2017 εγκρίναμε την πρόταση για την αναθεώρηση του ETS, του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών για την Αεροπορία. Όλες αυτές οι προστάσεις θα μας βάλουν στο σωστό δρόμο για να απαλλάξουμε την οικονομία μας από ανθρακούχες εκπομπές και να να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις των Παρισίων. Επίσης, θέλω ένα ηχηρό σήμα για τη δέσμευση και την προσήλωσή μας υπέρ της Συμφωνίας των Παρισίων και με την εφαρμογή του πακέτου για την ε, καθαρή ενέργεια και την πρόταση πρόοδο που θα κάνουμε δείχνουμε πόσο προσφυλής μας είναι η Συμφωνία των Παρισίων. Αυτά θα είναι όλα θετικά και για το πλανήτη και για την οικονομία μας. Θα τονώσουν την οικονομία, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και θα βοηθήσουν την ανάκαμψη της οικονομίας. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρώτη το 2017 και τώρα θα πρέπει να κρατήσουμε αμύωτες τι προσπάθειές μας και να συνεχίσουμε και στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 δεν ε, θα αφιστούμε προσπαθειών προκειμένου να παραμείνουν αμύωτες οι φιλοδοξίες μας και να τηρήσουμε τη συνοχή και το χρονοδιάγραμμά μας. Ε, Επίση, ε, ανταποκρινόμαστε στην έκκληση των Προέδρων των Τριοθεσμικών οργάνων το Δεκεμβρίου 2016 για να σημειώσουμε ουσιώδη πρόοδο και στα αποτελέσματα πριν τα τέλη του 2017. Η Εστονική Προεδρία έχει μια φιλόδοξη ατζέντα και επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα των ε, Συμβουλίων Υπουργών Ενέργειας για το δεύτερο εξάμεινο του 2017. Οπότε θέλουμε οι διοργανικές διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Ακούγεται φιλόδοξο, αλλά είναι ρεαλιστικό. Σε ό,τι αφορά τη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού, δείξαμε ότι είναι δυνατό μέσα σε 15 μήνες ε, να καταλήξουμε σε συμφωνία για τον κανονισμό SOS, IGA και τον κανονισμό πλαίσιο για την ε, επισήμανση στα ενεργειακά προϊόντα. Ήταν τριμερείς οι διάλογοι, ε, ήταν περίπλοκοι μάλλον οι τριμερείς διάλογοι, αλλά συνεχίζουμε με προσήλωση και πάθος ε, της προσπάθειας. Με τη, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους, Ένα σημαντικό τμήμα τη προπαρασκευαστικής μα εργασία είχε ολοκληρωθεί. Βέβαια, στις 31 Μαΐου υιοθετήσαμε τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα, το τελευταίο τμήμα των προτάσεων για την ενέργεια και θα συνεχίσουμε το έργο μας και σε άλλους τομείς τους επόμενους μήνες. Θα αναφερθώ στα εξή. Ω τμήμα της δέσμευσής μας για την ασφάλεια της, ε, της προμήθειας σε αέριο θα προτείνουμε ε, τροποποίηση της ε, συνθήκης για την ενεργειακή κοινότητα. Ε, επίσης ε, θα δημοσιεύσουμε τον τρίτο κατάλογο προ, ε, σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και με την ε, ανακοίνωση για 15% στόχο διασύνδεση για το 2030 και την αξιολόγηση του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και την αξιολόγηση ε, για τον κανονισμό για το Connecting Europe Ω τμήμα της ε, Ενεργειακής Ένωσης και του σχετικού πλαισίου θα ξεκινήσουμε την πλατφόρμα για περιοχές έντασης άνθρακα και περιοχές άνθρακα σε μετάβαση μαζί με το Φόρουμ για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά. Επίσης ε, θα εξετάσουμε τη, τα νομικά κοινά, κενά που υπάρχουν σε κάποιες ε, παράκτης, ε, παράκτης αγωγούς όπως είναι το Nord Stream. Αυτό είναι σημαντική προτεραιότητα. Επίσης μετά το πακέτο κινητικότητας της 31ης Μαΐου είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε ένα δεύτερο πακέτο πρωτοβουλειών μαζί με την νομοθεσία για τις διακοπές δεξιδίου του Άθρακα στα φορτηγά, ημιφορτηγά, ε, ε, πούλμαν, λεωφορεία και ταλίκες. Για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά ετοιμάζουμε νομοθεσία για την περίοδο μετά το 2020 με στόχους εμπορίας εκπομπών που θα ε, διευκολύνει τη μετάβαση προς χαμηλά και μηδενικής εκπομπής αυτοκίνητα. Επίσης εξετάζουμε τα, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών ε, και στόχο έχουμε να δώσουμε κίνητρα για τη δημιουργία ε, οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών. Επίσης θα εξετάσουμε ε, τι αντίκτυπο θα έχουν τέτοια οχήματα χαμηλών εκπομπών σε θέματα ηλεκτροδότησης, στις, στις θέσεις και στις δεξιότητες και μετά το 2020 με τις προδιαγραφές για τα αυτοκίνητα και τα μη φορτηγά θα επιταχύνουμε την εισαγωγή ε, στην αγορά τέτοιων αυτοκίνητων χαμηλών εκπομπών. Θα έχουμε όμως ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, με έμφαση όχι μόνο στην προσφορά αλλά και στη ζήτηση. Επίσης, ε, για να τεθούν στην αγορά τέτοια οχήματα, δεν αρκεί να έχουμε στόχου, γιατί η επιτυχία ηλεκτρικών ή άλλων οχημάτων χαμηλών εκπομπών ή μηδενικών εκπομπών θα εξαρτηθεί αφενό από τι διαθέσιμε υποδομέ για την επαναφόρτιση και από την άλλη από το πόσο γρήγορα θα είναι διαθέσιμες και σε προσιτές ανταγωνιστικές τιμές οι μπαταρίες οι σχετικές. Επίσης, ε, ανακοινώσαμε με το πακέτο για την κινητικότητα και κάποιες πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε την κατασκευή τέτοιων συνδεδεμένων και χαμηλών εκπομπών οχημάτων, αλλά και να αναπτύξουμε την κατασκευή μπαταριών νέας γενιάς στην Ευρώπη. Επίσης, με την νομοθεσία για το διοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να εναρμονιστούμε και με την παγκόσμια διαδικασία και να έχουμε πολύ ρεαλιστικούς ε, και σωστούς στόχους για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα από τα καυσαέρια. Επίσης, ε, θέλουμε τέτοιες οριακές τιμές ε, WLTP να είναι ρεαλιστικές, κατάλληλες για το σκοπό που εξυπηρετούν και να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της πραγματικής οδήγησης. Επίσης, για τα βαρέα οχήματα και τις εκπομπές τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε την πρόθεσή της να προτείνει προδιαγραφέ εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για το πρώτο εξάμεινο του 2018. Το αναλυτικό έργο για κάποιε επιλογές σχεδιασμού για τέτοιε προδιαγραφέ βαρέων οχημάτων συνεχίζεται αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να είμαι σαφή. Η πρότασή μα δεν θα είναι μια πιστή αντιγραφή απλώς προηγούμενων λύσεων για άλλου για για άλλους Θα στηριχθεί σε μια άρτια και εμπεριστατωμένη μελέτη επιπτώσεων που θα καταλήξει στην πρόταση μιας λύσης που θα είναι κατάλληλη για την αγορά μας, για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας και για να τηρήσουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς μας στόχους. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις για, τις, για την υλοποίηση των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής Γιούνκερ και προσβλέπω σε αγαστή και στενή συνεργασία μεταξύ μας γιατί αυτό πραγματικά προσδοκούν οι πολίτες από εμά. Όπως βλέπετε, με το τελευταίο τμήμα του 2017 και σε αρχές του 2018 θα έχουμε επιτάπητος ε, όλες τις προτάσεις ε, με βάση το πρόγραμμά μας και θα μεταβιβάσουμε τον μπαλάκι στο δικό σας γήπεδο γιατί θα πρέπει από κοινού να ξεκινήσουμε φιλόδοξους τριμέρις διαλόγους ώστε να καταλήξουμε σε κατάλληλη νομοθεσία που θα πληρεί τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Βεβαίω, ε, θα αντιμετωπίσουμε πολύ υπεύθυνα ό,τι μας στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε του εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Πολ Ρούμπιχ από πλευρά του ΕΛΚ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σα. Ξέρουμε ότι το φθινόπωρο θα έχουμε πολλές προκλήσεις ενώπιόν μας, ιδιαίτερα για την ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε τους στόχους, αλλά και να τους εφαρμόσουμε. Στην πολιτική το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές εργαζόμεθα τιμωρητικά με δεσμευτικούς στόχους, και σε ένα βαθμό αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια με τους πολιτικούς. Η, διαδικασία του Brexit, συμμετοχή σε ευρωεκλογές στη Σλοβακία 13%. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, ο τρόπος ε, εργασίας ημών των πολιτικών ε, επιτυχάνει τους στόχους μας. Θα ήταν πολύ καλό να σκεφτούμε τι ενάυσματα μπορούμε να δώσουμε για τους πολίτες μας, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί τα προβλήματά μας. Για παράδειγμα, στις μεταφορές. Τις αναφέρατε. Γίνεται πολλή συζήτηση για τα οχήματα εσωτερικής καύσης, αν θα πρέπει να επιτρέπονται στο μέλλον. Οι πράσινοι για πρώτη φορά ε, υπέβαλαν την πρόταση ότι μέχρι το 2000, ε, συγγνώμη, μετά το 2030 δεν θα πρέπει να παράγεται κανένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Και βλέπουμε επίσης ότι για αυτή την ε, ηλεκτρονική κινητικότητα χρησιμοποιούμε μπαταρίες ιόντος ε, λιθίου που ορισμένε δεν επιτρέπεται να μπαίνουν πια σε αεροπλάνα γιατί παίρνουν φωτιά. Αλλά όπως συζητήσαμε σε ένα ηλεκτρικό όχημα θα έχουμε 400 κιλά από τέτοιε μπαταρίες. Και άμα πάρει φωτιά όπως έγινε με το αεροπλάνο πώ θα, θα σβήσει με τις παραδοσιακές ε, μεθόδους αν μπει σε ένα, σε πάρκινγκ και υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα με τέτοιες μπαταρίες, καταλαβαίνετε τι μπορεί να προκύψει. Ε, τώρα η πρόσφατα στο Λονδίνο κάει και ένας ουρανοξύστης. Τι θα κάνουμε, θα απαγορεύσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μπαίνουν σε αστικές περιοχές και να παρκάρουν σε υπόγεια πάρκινγκ. Τι στρατηγική θα υιοθετήσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το θέμα της συνεχούς οδήγησης, α, δηλαδή να επιτυγχάνουμε σταθερές ταχύτητες. Αυτό θα δώσει στον κλάδο τη δυνατότητα να ε, δημιουργήσει νέα προϊόντα, να υπάρχουν αισθητήρε που θα καθορίζουν μια σταθερή ταχύτητα, να μην χρειάζεται δηλαδή να σταματάει κανείς στα φανάρια. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ λιγότερα ε, ε, πολύ λιγότερο καουτσούκ που θα λιώνει στους δρόμους γιατί δεν χρειάζεται να φρενάρουν και αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και καθαρότερο περιβάλλον. Επίσης, καταναλώνουμε τρομερή ενέργεια που βλάπτει, με τρόπο που βλάπτει τον καταναλωτή και τους ε, κατοίκους των ε, αστικών κέντρων. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέες προδιαγραφές για τα καύσιμα. Χρειάζονται επενδύσεις γι' αυτό. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να μειώσουμε την ενέργεια που μπορεί να ε, αποθηκευθεί σε ένα όχημα και η πυκνότητα των μπαταριών θα παίξει μεγάλο ρόλο στο μέλλον. Και σας παρακαλώ στο ένα το πρόγραμμα πλαίσιο να είναι προτεραιότητα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Ο κύριος Νταν Μίκα για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, Καταρχάς, ε, σας ευχαριστώ που τηρήσατε την υπόσχεσή σας όταν ε, συναντήσατε τους συντονιστές και σας ζητήσαμε μία ταχεία διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, για τη χρηματοδότηση. Έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους ε, για τα διάφορα θέματα, είτε είναι ανανεώσιμοι, είτε είναι ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες. Και για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους χρειαζόμαστε περισσότερες πιστώσεις. Οπότε, το ερώτημά μου είναι το εξής. Κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού προτίθεστε να αγωνιστείτε για να έχουμε την αναγκαία χρηματοδότηση για να επιτύχουμε αυτούς, αυτούς τους τόσο φιλόδοξους στόχους. Και επιπλέον, θέλουμε τους πόλους να προωθήσουμε για την ενέργεια, για το φυσικό αέριο. Και εδώ θα χρειαστούν τρομερές επενδύσεις για να επιτύχουμε τους στόχους. Είναι ακριβή αυτή η πόλη. Και για να επιτύχουμε τους στόχους μας Α, χρειαζόμαστε χρηματοδότηση. Γιατί δεν μπορούμε να να αφαιθούμε μόνο ε, στους ε, παρόχους υπηρεσιών και όχι στους τελικούς χρήστες. Πρέπει να βασιστούμε και στους δύο. Τώρα, Επιμένω ε, στο θέμα των ε, ηλεκτρικών ε, οχημάτων. Δεν ανησυχώ τόσο πολύ για το τι μπαταρίε θα έχουν. Ωστόσο, πιστεύω ότι η Ένωση θα πρέπει να βρει μια λύση. Τι υλικά θα χρησιμοποιούμε στην μπαταρία. Τώρα υπολοιπόμεθα των ΗΠΑ και της Κίνας. Είμαστε στην τρίτη θέση. Αν περιμένουμε δεν θα πάρουμε καθόλου μετάλλιο. σε μεγάλο βαθμό ε, οι μεταφορές είναι ο χειρότερος κλάδος από πλευράς μόλυνσης. Όλο και αυξάνονται οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακος από τον τομέα αυτό και προσπαθούμε να βρούμε διάφορες λύσεις. Προσπαθούμε να επιβάλλουμε, για παράδειγμα, την υποχρέωση να υπάρχουν σταθμοί φόρτισης στο 10-20% των ε, θέσεων παρκαρίσματος των θέσεων στάθμευσης ε, στα πάρκινγκ. Αλλά τώρα όσοι θέλουν να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα ε, περιμένουν να έχουν και δυνατότητες ε, να τα φορτίζουν. Θα πρέπει να υπάρχουν και σε περιοχές κατοικίας. Στην χώρα μου μπορεί να έχει κανείς ε, να λάβει κανεί 10.000 ευρώ επιδότηση για να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορεί κανεί να το αγοράσει γιατί δεν θα έχει που να το φορτίσει, θα πρέπει να το κρατήσει στον καράζ. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει πολύ ριζική παρέμβαση πλευρά τη Κομισιόν γιατί όλα τα άλλα δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τοσενόφσκι, ECR, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που επισκεφτήκατε την Επιτροπή μας. Ακριβώς αυτή τη στιγμή που πραγματοποιείται έντονη συζήτηση σχετικά με το ενεργειακό πακέτο. Η συζήτηση αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Δύο ερωτήσεις έχω να σας θέσω. Καταρχάς, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για την αύξηση σε 45 40 ή 45% των στόχων που έχουν καθοριστεί ως προς την βιώσιμη ενέργεια. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα αλλάξει αυτό το οικονομικό μοντέλο πάνω στο οποίο είχαν βασιστεί τα σχέδια σας όσον αφορά την ενίσχυση των ε, δικτύων μετάδοσης, των δικτύων μεταφοράς ενέργειας. Δεν είναι εύκολη η συζήτηση αυτή, διότι ε, έχουν αλλάξει πολύ οι στόχοι. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι επίσης τεχνικής φύσης. Στη δέσμη μέτρων υπάρχει ένας νέος όρος, περιφερειακά μέτρα διαχείρισης, ε, που τώρα πια έχουν αρμοδιότητες που δεν βασίζονται όμως σε προτάσεις που θα υποβάλουν τα ίδια. Έχουμε δει όμως ότι επειδή τα δίκτυα μεταφοράς αλλάζουν γρήγορα λόγω ε, της αιωλικής ηλιακής ε, ενέργειας και των φωτοβολταϊκών, πώς ανταποκρίνονται οι εθνικοί ρυθμιστές σε αυτές τις αλλαγές. Η απέτηση να δημιουργηθούν περιφερειακά κέντρα απέτει πολλούς ειδικού. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να ασχολούνται με τα δίκτυα και όπως γνωρίζετε είναι Ε, δύσκολη η κατάρτιση ανθρώπων ε, για να ε, γίνουν εθνικοί ρυθμιστές. Αυτό απαιτεί χρόνια. Εσείς πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το νέο μέτρο, τα περιφερειακά κέντρα. Για μένα το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι συστάσεις θα είναι μη δεσμευτικές. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Η κυρία Μάισνερ από την Άλντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ σήμερα. Πράγματι, όπως είπατε, ε, όσον αφορά την Ενεργειακή Ένωση, μέχρι το τέλος της χρονιάς ε, θα έχουν τεθεί όλες οι νομοθεσίες επιτάπητος. Ε, θα πρέπει λοιπόν κατόπιν να εφαρμόσουμε τις πολιτικές και η εφαρμογή είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική όσο οι αποφάσεις. Χθε είχαμε έντονη συζήτηση σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση, η Επιτροπή Ήτρε μαζί με την Επιτροπή Ένβη. Όλοι θέλουν να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά σε πολλά σημεία δεν σημειώνουμε πρόοδο. Οι άνθρωποι ανυπομονούν. Εγώ είμαι Γερμανίδα και υπάρχει εκεί ένα πανό που λέει ναι ενεργειακή ένωση αλλά δεν ε, βλέπουμε πρόοδο. Τι γίνεται λοιπόν στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε δίκτυα. Πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα για την Ενεργειακή Ένωση και φυσικά είναι σωστό να, ε, συμμετέχει και, να συμμετέχουν και οι πολίτες, αλλά για παράδειγμα, έχει σταματήσει ένα πρόγραμμα αιωλικής ενέργειας ε, στον Βορρά ε, επειδή ε, δεν καταναλώνεται τοπικά η ενέργεια. Λογικά, είναι όμως να έχουμε αιωλική ενέργεια στον Βορρά, ηλιακή ενέργεια στον Νότο. Χρειαζόμαστε όμως τις απαραίτητες υποδομές. Πώς έχει η κατάσταση. Η άλλη με ερώτηση είναι πολύ σύντομη. Κατάλαβα σωστά ότι θεωρείτε ότι το Nord Stream 2 είναι καλό πρόγραμμα διότι είναι επίμαχο το θέμα. Επίσης, όσον αφορά τις μεταφορές, διότι είμαι μέλος και της Επιτροπής Μεταφορών, ε, βρίσκω σωστό ότι λέτε ότι πρέπει να ποντάρουμε στην ηλεκτροκινητικότητα. Ε, άλλες χώρες ε, ποντάρουν στο υδρογόνο. Πάντω έχουμε πρόταση από την προηγούμενη θητεία που αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται στη φάση εφαρμογής. Αλλά ούτε σε άλλε χώρε ούτε στη Γερμανία είναι όλα έτοιμα. Χρειαζόμαστε υποδομή, αυτό όμως σε πολλές περιπτώσεις ε, χρειάζεται κάποια χρόνια ακόμα. Θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη πέρα από το θέμα της ε, ενέργειας που συνδέεται και με τη βιομάζα και με άλλα υλικά που χρειαζόμαστε. Αυτό ισχύει και για τις αερομεταφορές. Είσαστε Ισπανός. Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Ε, και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μπορούμε να εξοικονομήσουμε εδώ ενέργεια. Ε, γνωρίζετε επίσης το θέμα του Γιβραλτάρ και θα βρεθεί ποτέ εκεί η διπλωματική λύση. Είναι πολύ δύσκολο. Να εξηγήσουμε στους πολίτες ε, ότι τα αεροπλάνα αναγκάζονται να κάνουν ζιγ-ζακ ε, και ότι δεν μπορούν να πετούν σε ευθείες γραμμές. Είσαστε σε θέση να επηρεάσετε την ε, κυβέρνηση στην πατρίδα σας ώστε να προοδεύσουμε όσον αφορά το θέμα της, ηλεκτρικής, της ενεργειακής απόδοσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρίβαση από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κανιέτε που ήρθατε, γιατί έχετε σημαντικότατες ε, ευθύνες. Θα θέλουμε να ευοδοθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, ή την ενεργειακή απόδοση και συμβατές ε, με τη διακήρυξη του Παρισιού θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι γιατί οι τελευταίες ερευνές δείχνουν ότι ναι μεν είμαστε 27% αν μείνουμε στο 27% για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή απόδοση, δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας από τη Συμφωνία του Παρισιού. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το μεθάνιο. Όταν διαβάζουμε τις εκθέσεις, διαπιστώνουμε ότι το μεθάνιο είναι από τα πιο επιζήμια αέρια του θερμοκηπίου και μάλιστα και βραχυπρόθεσμα επιζήμιο. Και μια, έχουμε, και έχουμε στόχους για το 2050, μέχρι το 2050, σε πολύ μακρινό χρονικό ορίζοντα. Ερωτώ, μήπω θα μπορούσαμε να έχουμε ειδική στρατηγική για το μεθάνιο, γιατί ένα τόνο μεθανίου ε, αντιστοιχεί σε 21, 21 τόνους διοξίδιο του άνθρακα για 100. Αν όμως το δούμε βραχυπρόθεσμα σε 5 χρόνια, είναι πολλαπλάσια η αρνητική επιρροή. Οπότε, αν έχουμε ειδική στρατηγική για το μεθάνιο, θα καταφέρουμε πιο εύκολα να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Πότε πρόκειται να μας υποβάλλετε λοιπόν πρόταση στρατηγικής για το μεθάνιο γιατί έτσι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τις συμφωνίες του Παρισιού και σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Είπατε επίσης ότι θέλουμε 27% μερίδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με βάση μια μελέτη επιπτώσεων ε, για το κόστος που ήταν υπερτιμημένο. Ενώ σήμερα όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το πραγματικό κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολύ πιο μικρό, πολύ πιο χαμηλό Ερωτώ λοιπόν κυρία Κανιέτε, πότε θα μας υποβάλλετε μια νέα αξιολόγηση των στόχων των ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό και όχι το υπερτιμημένο κόστος. Αυτό θα πρέπει να ζητήσετε από τις υπηρεσίες σας, μια ενημερωμένη μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη το πραγματικό κόστος, ώστε να είμαστε πιο φιλόδοξοι για τις ΑΠΕ, την ενεργειακή απόδοση, αλλά και τη μείωση της κατανάλωσης. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδυάσουμε για να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας στη Συμφωνία στο Παρίσιου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπενίτο Θηλουάγα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, ολοκληρώθηκαν οι δημόσιες διαβουλεύσεις για τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά και τις διασυνδέσεις σε υποδομές φυσικού αερίου. Και για τις τελευταίες υποδομές θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί αυτό που επιχειρείται είναι να δοθούν δημόσια κονδύλια στην πρόθεση ε, ορυκτού αερίου με αντί να επενδύουμε κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ενεργειακή απόδοση με δημόσια κονδύλια. Αυτό τι ενέργεια έχει χαρακτηριστικά ε, περιβαλλοντικού εγκλήματος. 86 το δυναμικό ε, υπερθέρμανση του μεθανίου είναι 86 φορές μεγαλύτερο από το δυναμικό του διοξιδίου του άνθρακα. Αν διαβάσετε μελέτες του Πανεπιστημίου της Κορνοάλης, διαπιστώνετε ότι συνδέεται η ιδέα της εκπομπές μεθανίου με τις προσπάθειες εξόριξης ε, φυσικού αερίου. Οπότε αν δώσουμε έμφαση σε τέτοιο αέριο θα αυξήσουμε και τις εκπομπές μεθανίου που είναι το πιο επιζήμιο αέριο του θερμοκηπίου. Επίσης, σε σχέση με τα έγγραφα του Παναμά, μας είχατε πει σε μία ακρόση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ότι δεν έχετε καμία άμεση σχέση με τις επιχειρήσεις που εμφανίζονται στα έγγραφα του Παναμά. Τις τελευταίες όμως εβδομάδες διαπιστώσαμε ότι η ΟΛΑΦ σας έχει στο στόχαστρο των ερευνών της. Και μάλιστα πολλοί έχουν παραιτηθεί για διασυνδέσεις με τα, με τα έγγραφα του Παναμά. Ο πρώην Υπουργός Όρια, ο Διασαγγελέας Βόρης, παρόλο που στην αρχή ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία σχέση και τελικά χρειάστηκε να παραιτηθούν όταν αποδείχθηκε η άμεση σχέση τους. Μήπω θα μα εμφανιστείτε κι εσείς ε, τελευταία στιγμή να έχετε άμεση σχέση και θα αναγκαστείτε να παρατηθείτε. Η, η υπογραφή που έχει βάλει ένα συγγενή σα αν εμφανιστεί στη διακήρυξη, στη δήλωση ε, σύγκρουση συμφερόντων που υποχρεωθήκατε να υπογράψετε για να αναλάβετε ως επίτροπος, δεν θα πρέπει να αναγκάσει και εσάς σε παρέτηση όπως και άλλους συναδέλφους σας. Ευχαριστώ. Ah, wonderful. Thank you. Okay. First. Well, thank you all of you for your questions. Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις του κυρίου Ρούμπιχ. Για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος από τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά θα πρέπει να είναι πολύ περίπλοκο αυτό που κάνουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ρόλο παίζει στις θέσεις εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τους κατασκευαστές αλλά και όλους τους υπεργολάβους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Παίζει μεγάλο ρόλο στην βιομηχανική παραγωγή και στις εξαγωγές της Ένωσης αυτός ο κλάδος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά και με ολιστική προσέγγιση πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα απλώ να υπάρχουν προδιαγραφές, είναι πώς θα χειριστούμε την κυκλοφορία, πώς θα οργανώσουμε τις ροές οχημάτων στις πόλεις, πώς θα οργανώσουμε τη μετάβαση στις μεταφορές χωρίς παραγωγή οξυδίων του άνθρακα είναι μια μετάβαση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε 10 χρόνια θα καταργήσουμε τις μηχανές εσωτερική καύση. Γιατί μπορούμε να βελτιώσουμε κατά πολύ ακόμη αυτούς τους κινητήρες. Έχουμε συζητήσει πολλές τεχνολογίες για να δούμε σε τι βαθμό θα βελτιωθεί η κατάσταση, πόσο θα βελτιωθεί η απόδοση των κινητήρων σε σχέση με το κόστος. Αλλά για να επιτύχουμε φιλόδοξους στόχους μείωσης ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, θα πρέπει να υπάρξει πολύ περισσότερη ηλεκτρική κινητικότητα. Οι κατασκευαστές για να κατασκευάσουν τέτοια αυτοκίνητα χρειάζονται ζήτηση. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ότι θα να επιβάλλουμε στους κατασκευαστές ότι θα παράγεται 20 εκατομμύρια τέτοια αυτοκίνητα, ακόμη και αν χάνεται 3.000 ανά αυτοκίνητο. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε ζήτηση. Και για να δημιουργήσουμε ζήτηση θέλουμε σημεία φόρτισης και θέλουμε καλύτερες μπαταρίες. Αυτές είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Η Κομισιόν λοιπόν δεν μπορεί να πει «Α, ας θέσουμε ένα στόχο» να πάει στα τόσα γραμμάρια. Όχι. Πρέπει να μπουν οχήματα χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών στην αγορά. Πρέπει να υπάρχουν. Αλλά πρέπει να ε, καταστήσουμε δυνατή την κυκλοφορία τους. Άρα χρειαζόμαστε σταθμούς φόρτιση, είτε πρόκειται για, για ε, μπαταρίες υδρογόνου, είτε πρόκειται για ηλεκτρικές μπαταρίες, είτε πρόκειται και για ε, σταθμούς φόρτισης υψηλής ταχύτητας και χαμηλής ταχύτητας. Και επίσης, αν δείτε τι λέει η οδηγία μας για την ενεργειακή απόδοση, Έχουμε πει ότι τα νέα κτίρια πρέπει να έχουν προκαταρκτική παρουσία των καλωδίων. Να υπάρχουν τα καλώδια, ε, να υπάρχουν τα καλώδια που κοστίζουν για παράδειγμα 300 ευρώ και μετά αν θέλεις να βάλεις εκεί του, τα σημεία φόρτισης να τα βάλεις τα πληρώς 2.000. Και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει επίσης στα δημόσια πάρκινγκ ένα ε, σταθμό φόρτισης ένα σημείο φόρτισης ανά 10, σημεία, ανά 10 χώρους ε, στάθμευσης. Ανά 10 θέσεις στάθμευσης. Θα πρέπει και στα πάρκινγκ, στα σούπερ μάρκετ, όπου είναι δυνατόν, στα μεγάλα κέντρα αναψυχής, ε, στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όπου υπάρχουν τέτοια πάρκινγκ πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες φόρτισης και ε, πάνω στις κύριες αρτηρίες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα βασικό σχέδιο για να ε, στηρίξουμε την κυκλοφορία των οχημάτων χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να χάσουμε τη μάχη της μπαταρίας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις υπάρχουσες πιστώσεις από το Horizon 2020, από οπουδήποτε, για να κατασκευάσουμε μπαταρίες νέας γενιάς. Να κάνουμε ρηξικέλευθες ε, ανακαλύψεις για τα θέματα αυτά και να φτιάξουμε και τα εργοστάσια που θα παράγουν αυτές τις μπαταρίες εδώ στην Ένωση. Και αυτό είναι περίπλοκο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει ο διάλογος με τους κατασκευαστές, ποια στήριξη θα τους δώσουμε για να αναπτύξουν αυτές τις νέες μπαταρίες. Δεν πρέπει να χάσουμε τη μάχη της μπαταρίας, της μπαταρίας της νέας γενιάς. Ήδη και τώρα το, με τα ιόντα λιθίου είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζονται τεράστιες ε, εγκαταστάσεις για να κατασκευαστούν. Τώρα δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε, αλλά πρέπει να ανταγωνιστούμε στις μπαταρίες της επόμενης γενιάς. Και αυτό κύριε Ρούμπιχ είναι πολύ περιπλοκό. Γιατί πρέπει να επιτύχουμε και τους κλιματικούς μας στόχους, αλλά για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει οι αυτοκινητοβιομηχανίες να γίνουν πολύ καλύτερες. Πρέπει λοιπόν κάτι να αλλάξει και πρέπει να προβλέψουμε. Οι κινητήρες εσωτερικής καύση θα παραμείνουν. Ακόμη μπορούν να βελτιωθούν, αλλά φυσικά θα μειώνεται η χρήση τους. Γιατί θα αυξάνεται η χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων και των οχημάτων χωρί οδηγό. Και τι έχει να γίνει με τι δεξιότητε. Οι εργάτε τώρα στα εργοστάσια ε, είναι ειδικευμένοι για να κατασκευάζουν κινητήρια εσωτερική καύση. Δεν έχουν τι αναγκαίε δεξιότητε για να λειτουργούν μπροστά σε υπολογιστέ για να παράγονται τα νέα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσουμε και το εργατικό δυναμικό. Να το επανεκπαιδεύσουμε. Α, αυτή είναι η πρόκληση μπροστά μα. Πρέπει να κάνουμε μια πρόταση που να είναι πολύ σωστά ισορροπημένη. Δύο χρόνια χωρίς να δρώ βεβαιασμένα, προσπαθώ να καταλήξω σε λύση για το θέμα αυτό γιατί είναι πολύ περίπλοκο. Όλες οι προτάσεις ε, που έχουμε υποβάλει είναι πάντα βεβαίως ε, ε, περίπλοκες, αλλά αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Τώρα, Νίκα, πού είναι ο Νίκα. λοιπόν. Α, διασυνδέσεις και χρηματοδότηση αυτών. Θα συζητήσουμε τις νέες ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Και φυσικά η κλιματική ε, αλλαγή είναι 20% σε όλα. Θα υπάρχει 20% και από τα διαδροτικά ταμεία και το σχέδιο Juncker θα χρηματοδοτεί όλο και περισσότερα προγράμματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Στην αρχή υπήρχαν δυσχέρειε λόγω των προβλημάτων ενεργειακή απόδοση. Ήταν δύσκολο να υπάρχουν μεγάλα προγράμματα για την ενεργειακή απόδοση, αλλά τώρα έχουμε περισσότερε δυνατότητε. Θα έχουμε και την πρωτοβουλία για τα κτίρια, θα έχουμε και το ΣΕΦ, αλλά στο τέλο είναι σαφέ, δηλαδή στη τελευταία ανάλυση, είναι σαφέ ότι η δημόσια, η δημόσια χρηματοδότηση θα είναι ένα μικρό τμήμα. Για να υπάρξει η σωστή χρηματοδότηση πρέπει να υπάρχει μια αγορά γιατί χρειαζόμαστε ιδιωτική χρηματοδότηση για τις ανανεώσιμες και ένα αριθμιστικό πλαίσιο που να τους υπόσχεται σταθερότητα, μακροπρόθεσμη, ούτως ώστε οι επενδυτές να μπορούν να πούνε βεβαίως καταλαβαίνουμε για τα επόμενα χρόνια ξέρουμε ότι θα υπάρξουν ε, προγράμματα κλιματικής δράσης από τις κυβερνήσεις υπάρχει προβλεψιμότητα. Και φυσικά θα πρέπει να αλλάξουμε κάποιους κανόνες για τα συμβόλαια ενεργειακής απόδοσης. Να είναι απλούστερα, να μπορεί η δημόσια δίκηση να τα προωθήσει. Κοζανόφσκι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα. Τα ΡΟΚ. Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι πολύ πιο διασυνδεμένο από το παρελθόν γιατί υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ανανεωσίμων στο ενεργειακό μείγμα. Οπότε τα συστήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε εθνικό επίπεδο, αλλά περιφερειακό. Στο παρελθόν ήταν εθελούσια συνεργασία. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν έχουν πολλές αρμοδιότητες ε, αυτά τα ροκ. Δεν αντικαθιστούν τους άλλους φορείς ε, λειτουργίας του δικτύου. Μόνο εάν άλλοι φορείς δεν μπορούν να φτάσουν σε αποτελεσματική λύση παρεμβαίνουν. Οι λειτουργίες λοιπόν αυτών των ΡΟΚ θα ε, γίνουν πολύ πιο αποφασιστικές στο μέλλον για να υπάρχει σωστή λειτουργία του συστήματος. Ε, ορισμένοι θεωρούσαν ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Αυτά τα ροκ θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνα αν υπήρχε τρομερή αμέλεια και θα έπρεπε να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη. Και αυτό είναι παράλληλο με αυτό που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Θα έχουν λοιπόν τις αναγκαίες ικανότητες και θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Τέθηκε και μία ερώτηση από τον κύριο Τουσενόφσκι σχετικά με την ε, αύξηση των στόχων. Θεωρήσαμε ότι η καλύτερη αναλογία κόστους όφελους ε, μπορούσε να επιτευχθεί με 27% ε, ενεργειακή απόδοση και 30% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Κοινοβούλιο μπορεί να έχει άλλο επίπεδο φιλοδοξίας, ε, μπορεί να λαμβάνουμε νέα στοιχεία τα οποία πρέπει να εξετάσουμε όσον αφορά την κυρία Ριβαζή. Όταν λάβαμε υπόψη μας τις τιμές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, δεν ήταν οι τελευταίες διαθέσιμες τιμές. Και στην μελέτη αντικτύπου αξιολογούμε διάφορα σενάρια. Θα γίνει αυτή η αξιολόγηση, αλλά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι αυτή που είναι. Θα εξετάσουμε τις συνέπειες ε, αλλαγής των στόχων και θα επανέλθουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τη στείλουμε στον πρόεδρο της Επιτροπής σας, ώστε οι ευρωβουλευτές να μπορούν να τη διαβάσουν. Όσον αφορά τις διασυνδέσεις, αυτό είναι πάντα δύσκολο θέμα, διότι πρέπει να περνάμε τα σύνορα, αλλά μερικές φορές υπάρχουν και προβλήματα εντός της ίδιας χώρας, το οποίο είναι λιγότερο κατανόητο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες ε, Εάν προσπαθούμε να περάσουμε τα πυρηναία, πρέπει να εξετάσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ε, μπορεί να χρειαστεί να δουλέψουμε υπογείως. Ε, και γι' αυτό τώρα η διασύνδεση Γαλλίας και Ισπανίας γίνεται με τον τρόπο που γίνεται. Στη Βαλτική επίσης, η διασύνδεση των χωρών της Βαλτικής με το υπηρετικό δίκτυο θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα γίνει μέσω Πολωνίας ή μέσω των βορείων χωρών. Δεν είναι εύκολες αυτές οι διασυνδέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως πιστεύει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας. Θέλουμε λοιπόν να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι κάτι τέτοιο είναι θετικό για την εσωτερική αγορά και θα επιτρέψει περισσότερη ανάπτυξη. Θα υποβάλουμε λοιπόν έκθεση σχετικά με το πώς μπορούμε να πετύχουμε ε, τον στόχο του 15% και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, το θέμα του Γιβραλτάρ είναι πάρα πολύ δύσκολο, τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει και δεν γνωρίζω τι θα γίνει ένας ταπεινός επίτροπος είμαι, δεν νομίζω ότι έχω τη δυνατότητα να αλλάξω τις θέσεις της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε λιγότερες εκπομπές και λιγότερη χρήση καυσίμων. Σημειώνω πάντως την παρατήρησή σας. Κατόπιν είχαμε την ερώτηση του κυρίου Μπενίτο Θηλουάγκα. Είναι σαφές ότι στο παρελθόν, όταν είχαμε τη διακοπή παραχής αερίου του 2009, που σταμάτησε η τροφοδότηση από την Ουκρανία, ξεκινήσαμε ένα stress test για να δούμε τι επενδύσεις θα μπορούσαν να γίνουν με ευρωπαϊκό χρήμα για να μπορούμε να έχουμε ασφάλεια τροφοδοσίας. Στηρίξαμε λοιπόν διάφορα προγράμματα για να το πετύχουμε αυτό. Πάντως γίνεται όλο και πιο σημαντική η ισορροπία ανάμεσα στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, διότι χρειαζόμαστε τεράστιες επενδύσεις ε, στο ε, ε, ηλεκτρικό ρεύμα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο φυσικό αέριο κλπ. Τώρα λοιπόν θα αλλάξει η κατάσταση. Και θα δούμε μεγάλες αλλαγές στα προγράμματα του μέλλοντος. Πάντως, στο παρελθόν ήταν σαφής η κατάσταση, είχαμε μεγάλη κρίση το 2009 και έπρεπε να αξιολογήσουμε τα διάφορα προγράμματα, να ε, δημιουργήσουμε τον νότιο διάδρομο, και να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις άλλες χώρες. Και σας παραπέμπω και στις παρατηρήσεις μου σε άλλη επιτροπή ότι έχω σεβαστεί απολύτως τον κώδικα διοντολογίας των επιτρόπων. Συγγνώμη κύριε Κανιέτε. Δεν μου είπατε τίποτα για το μεθάνιο. Α, ναι, για το μεθάνιο. Όσον αφορά το μεθάνιο, ε, στον κανονισμό για τον επιμερισμό της προσπάθειας, Ένας από τους τομείς που αναφέρονται είναι η γεωργία, όπου είναι πολύ σημαντικές οι εκπομπές μεθανίου. Τα κράτη-μέλη λοιπόν στα σχέδια δράσης θα πρέπει να αναφέρουν τι κάνουν στους διάφορους τομείς ε, συμπεριλαμβανομένες της γεωργίας και τι κάνουν για να μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει αν οι προσπάθειές τους αρκούν. Αυτή τη στιγμή δεν ε, εκπονούμε συγκεκριμένη στρατηγική για το μεθάνιο. τουλάχιστον από πλευρά των υπηρεσιών μου. Αλλά ε, στα σχέδια δράσης για το κλίμα θα εξετάσουμε τι ε, συμβαίνει με το μεθάνιο και θα εξετάσω και όλα σε αν άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουν κάτι για το θέμα αυτό. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. αρκετά μακροσκελή ο κατάλογος των ομιλητών. Παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το δίλεπτο. Ο κύριος Ρόιλ. Δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, όσον αφορά ε, το νέο υπολογισμό των στόχων για τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Πώς κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα συγκεκριμένα νούμερα τυχαία ή υπάρχουν ε, συγκεκριμένες αιτίες. Διότι το Κοινοβούλιο ε, έχει άλλα νούμερα. Πώς έχετε καταλήξει λοιπόν ε, στους δικούς σας στόχους. Επίσης ε, αναφέρεστε στα κτίρια και το, τους σταθμούς φόρτισης. Εάν όμως το κάνουμε αυτό στα σούπερ όπου ε, συνήθως ε, μένει κανείς σε 30 λεπτά χρειαζόμαστε ε, σταθμούς γρήγορης φόρτισης. Οι σταθμοί αυτοί στοιχίζουν 25 με 30.000 ευρώ ανά σταθμό. Δεν μου φαίνεται ότι έχει κάποια λογική αυτό και εάν δημιουργήσουμε σταθμούς γρήγορης φόρτισης και σε κάθε σούπερ μάρκετ έχουμε πέντε τέτοιους σταθμούς, αυτοί θα στοιχήσουν σε ηλεκτρικό όσο καταναλώνει το σούπερ μάρκετ συνολικά. Πιστεύετε ότι αυτή είναι καλή λύση. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρος μας, ο κύριος Κόχλιτσεκ. Σας ευχαριστώ. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν, αργή φόρτιση. Χρειάζονται ειδικοί σταθμοί. Για την ταχεία φόρτιση ε, χρειάζονται 64 αμπέρ, στην αργία 32 αμπέρ. Δεν το έχουμε όμως αυτό σε όλα τα σπίτια, δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες και θα δημιουργήσουμε προβλήματα στα ηλεκτρικά οχήματα. Επίσης, το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη για το φυσικό αέριο έχουμε οδηγία για τη διασύνδεση βορρά και νότου. Υπάρχει δυνατότητα όντως να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο της διασύνδεσης βορρά και νότου. Άλλο θέμα. Στόχοι εκπομπών. Θα πρέπει να έχουμε στόχους εκπομπών όχι μόνο για το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά και για άλλα καυσαέρια. Υδρογονάνθρακες, αιωρούμενα σωματίδια, PM10 και ούτω καθεξής. Επίσης, τι γίνεται με τις μπαταρίες υδρογόνου, δεν είπατε τίποτα. Σε νέα μεγάλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται δοκιμές με λεωφορεία που χρησιμοποιούν ως καύσιμο υδρογόνο. Ενώ ταυτόχρονα κάποια εργοστάσια θα κλείσουν επειδή δεν υπάρχει ζήτηση, γιατί να μην τα ανακυκλώσουμε να παράγουν ε, στοιχεία ε, υδρογόνου, κύτταρα υδρογόνου που να χρησιμοποιεί το για την μηχανοκίνηση. Επίσης, φωτοβολταϊκά στοιχεία. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί δεν έχουμε πάντα ηλιοφάνεια για να συλλέγουμε τον ήλιο στα φωτοβολταϊκά. Το ίδιο ισχύει και για την αιωλική ενέργεια. Επίσης, λίγες χώρες στην Ευρώπη έχουν υποδομή Υψηλή τάση. Ε, και αυτό γίνεται θελοντικά. Τώρα ένα ε, άσχετο γραφειοκράτη, θα θέτει του κανόνε, αυτό θα είναι καταστροφή και θα διαλύσει το δίκτυο. Επίση για το μεθάνιο. Τι θα κάνετε, θα απαγορεύσετε τι αγελάδε, να μετεωρίζονται για να μην παράγουν ε, μεθάνιο. Αυτό είναι παράλογο. Να το λάβουμε υπόψη και επίσης να προσέξουμε την εξηγέση των υδάτων, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι για το μεθάνιο. Ε, υπερβήκατε το δίλεπτο, κύριε Κόχλιτσεκ. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες είναι ο επόμενος μας ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τις προάλλες ακούσαμε για την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένε Πολιτείε από τη Συμφωνία του Παρισιού. Αυτή η απειλή που δεν είναι πια απειλή, έγινε πραγματικότητα, δίνει μια ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πρωτοστατήσει, να αναλάβει ακόμη μεγαλύτερο ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια απαλλαγή τη οικονομίας από τις ανθρακούχε εκπομπές και να προωθήσει καθαρές ενέργειες, μεταξύ άλλων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα, κύριε Επίτροπε, επαναλάβατε την ανάγκη το χειμερινό πακέτο να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό και χαράξετε ένα μονοπάτι με νέους στόχους που αφορούν τη συνέχιση του γενικού μας στόχου που είναι η απαλλαγή της ε, οικονομίας μας από τον άνθρακα μέχρι το 2050. Εγώ στενίζω με το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνώ με την αντίδραση που είχατε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η G7 απέναντι στην απειλή του ε, Τραμπ που τελικά πραγματοποιήθηκε. Αν δεν δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν δεν επισπεύσουμε τη διαδικασία σε κάποιους στόχους, για παράδειγμα για τις μπαταρίες, για την ηλεκτροκίνηση και ούτω καθεξής, τότε δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε τις αγαθές μας προθέσεις και τους αξιέπαινους στόχους μας. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εσά, κύριε Επίτροπε, να σταθείτε στο πλευρό μας ώστε να υλοποιήσουμε πιο φιλόδοξους στόχους από αυτούς που θέσαμε αρχικά. σε σχέση με μελέτες που είχαν γίνει και πριν την COP21 του Παρισιού. Στηρίξτε μας, ε, γιατί είναι σημαντικό σήμερα να γίνουμε ακόμη πιο φιλόδοξοι σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο, την τήρηση της Συμφωνίας του Παρισιού. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ονκέλη είναι ο επόμενος μου ομιλητής στον κατάλογο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, παρουσία Δεν ήμουν από νωρίς, γιατί ήμουν σε ένα πρόγραμμα εργασία για την τοπική διάσταση της ενεργειακής μετάβασης. Τι μπορείτε να κάνετε και εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς, ώστε να αναμειχθεί και να αναμειχθούν και οι τοπικοί περιφερειακοί παράγοντες και να μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε τους στόχους του Παρισιού και να γίνουμε παγκόσμιοι ηγέτες σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την ενεργό ανάμειξη των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων. Είπατε ότι θα αναθεωρηθούν ε, οι στόχοι με βάση τις πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες. Είπατε όμως ότι σε μερικές πτυχές θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ακόμα και τα χρονοδιαγράμματα που θέσαμε όμως μήπως παρά είναι γρήγορα. Μήπως... Ε, σπέβδουμε υπερβολικά και δεν δίνουμε αρκετό χρόνο στι τοπικέ και περιφερειακές αρχέ και στι εθνικέ κυβερνήσει και στους ενδιαφερομένους να αναμειχθούν και αυτοί ενεργά. Δεν είναι καλύτερο αυτό από το να βιαστούμε χωρίς λόγο με κίνδυνο να οδηγηθούμε σε λάθος μέτρα. Επίσης, αναφερθήκατε στα εθνικά σχέδια δράση. Και, αλλά έχουμε και ένα γενικό κοινοτικό στόχο πέραν των εθνικών. Πώς ε, θα εξασφαλίσουμε την σύγκριση, τη συγκρισιμότητα αυτών των στόχων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτά. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι για τις προσπάθειές σας. Και τώρα, ο κύριος Ζουρίνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Το τελευταίο διήμερο στις Βρυξέλλες είχαμε τους πιο θερμές ημέρες της δεκαετίας. Και στην πατρίδα μου ο συνδυασμός ε, ψηλόθερμοκρασιών θερμοκρασιών ε, και μεγάλης υγρασίας μας οδήγησαν σε μια τεράστια καταστροφή με δεκάδες νεκρούς με τις πυρκαγιές. Και σε αυτό το υπόβαθρο η Αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Συμφωνία του Παρισιού. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσει τους στόχους ε, και τις δεσμεύσεις της από τη Συμφωνία του Παρισιού. Και μάλιστα ο κανονισμός για την ενεργειακή διακυβέρνηση, στον οποίο είμαι σκιώδης ηγετής, θα είναι πραγματικά η λιδία για μας. Και είναι σημαντικό αυτός ο γνώμονας ε, της ε, διακυβέρνησης να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη Συμφωνία του Παρισιού. Αν δεν υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση με το υπόδειγμα της ενεργειακής ε, διακυβέρνησης και της συμφωνία του Παρισιού, θα χάσουμε κάθε αξιοπιστία και κύρος στα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό για τον κόσμο να δείξουμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά τον αγώνα μας για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και θεωρώ ότι και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ακολουθήσει αυτή την άγουσα. Ερωτώ λοιπόν, θα μας συμπαρασταθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει συμμαχός μας, ώστε η ενεργειακή διακυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις δεσμεύσεις μας που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι δύο μου μένουν στο κατάλογο. Ο Ζάνθος Τούρμες. Ευχαριστώ, Ζέρζη. Κύριε Επίτροπε. Η Λιδία για το πόσο η Ευρώπη δεσμεύεται για όλα αυτά. Έλεγα λοιπόν ότι το αποφασιστικό θα το έχουμε τη Δευτέρα όταν ε, θα συζητήσουν οι Υπουργοί την νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση για τα κτίρια. Την τρίτη το πρωί κάνετε μια πολύ ενθουσιώδη ομιλία. Από ό,τι κατάλαβα έχουμε ένα νέο κείμενο τη Μαντέζικη Προεδρία. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία να υπάρξει συμφωνία τη Δευτέρα. Αλλά μια μεγάλη χώρα, η Ισπανία, δεν συμφωνεί του παρόντος. Συζήτησα με τον Ισπανό Υπουργό και μου είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ισπανία είναι οι λογιστικοί κανόνες, Eurostat. Μπορείτε να με βεβαιώσετε ότι θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα με αυτούς τους ε, κανόνες. Συμμετείχα με το Σόν σε αυτό το πρωινό εργασίας. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα για τις πόλεις για την ε, χρηματοδότηση από τρίτους ε, της ενεργειακή απόδοσης είναι αυτή η λογιστική κανόνα. Επίσης, χρειαζόμαστε δύο δίκτυα τώρα. Ισπανία, Πορτογαλία προς Γαλλία, το καλώδιο από τη Βισκάγια, από την, ε, ναι, από την από το Βυσκαϊκό κόλπο, ναι. Και το άλλο από την Γαλλία προς την Ιρλανδία. Και από ό,τι μου είπαν, η ανάλυση για το, τη σχέση κόστους-οφέλους είναι αρνητική για αυτά τα δύο δίκτυα, για αυτά τα δύο συστήματα καλωδίων. Και ενώ θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν από το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, υπάρχει κάποια ασάφεια φαίνεται, εάν αυτές οι αρνητικές αναλύσεις σημαίνουν ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν ή όχι. Δεν είναι παράλογο αυτό. Δημιουργήσαμε αυτό το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη για να βοηθήσουμε την Ισπανία και την Πορτογαλία <clears throat> να έχουν πρόσβαση στη Γαλλία και να διατηρηθεί η σύνδεση μεταξύ ε, Ιρλανδίας και Ευρώπης τώρα που η Βρετανία έχει σαλπάρει για το Τέξας. Ε, δεν θα πρέπει να ε, δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα των αναλύσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορώ και εγώ να πάρω το λόγο τώρα ως τελευταίος. Κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου αφορά το νέο σχεδιασμό των αγορών για το φυσικό αέριο. Γιατί χρειαζόμαστε συμβατότητα και νομίζω ότι τέλος του χρόνου και αρχές του επόμενου χρόνου θα έχουμε τις προτάσεις για αυτό το θέμα. Έχουμε επανειλημμένα συζητήσει το θέμα του Nord Stream 2 όπου είπατε ότι θέλετε να συζητήσετε ένα νέο νομικό πλαίσιο για το βαλτικό τμήμα αυτού του Nord Stream 2. Οπότε η ερώτηση. Πότε θα ήταν δυνατόν έστω και με βάση την εμπιστευτικότητα θα μπορούσατε να μας δώσετε πρόσβαση στα νομικά επιχειρήματα της Επιτροπής που ισχυρίζονται ότι υπάρχει ένα νομικό κενό και δεν μπορεί να καλυφθεί πύρο στο Nord Stream 2 από το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Και νομίζω ότι αν υπάρχει συμφωνία επί ενός νέου νομικού πλαισίου που τελικά είναι πιο αποδυναμωμένη από αυτή που προβλέπει το τρίτο ενεργειακό πακέτο αυτό δεν σημαίνει ότι δίδεται ένα θέμα το ένα συγγνώμη, μία, ένα θέμητο προνόμιο στο Nord Stream 2. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το τρίτο είναι πακέτο. Και το Nord Stream 2 πρέπει να καλύπτονται απόλυτα. Δηλαδή, ιδιαίτερα το τμήμα της Βαλτικής. Γιατί ορισμένα ε, τμήματα περνάνε από τα ύδατα κάποιων κρατών μελών της Ένωσης. Αυτό το θέμα, συγκρισιμότητα, συμβατότητα μάλλον των δύο αγορών. Και τρίτο ενεργειακό πακέτο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Όχι. Παρακαλώ. Ας ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Χρειαστήκαμε πολύ συζήτηση για να διαπιστώσουμε αν το τρίτο ενεργειακό πακέτο θα ισχύει και για τα υπεράκτια πάρκα ή όχι. Διότι εάν ε, μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την αποσύνδεση των δικτύων και όλους τους διάφορους κανόνες αλλά τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό ήταν μεικτό. Διότι οι μέτοχοι ήταν αφενός η Gazprom και αφετέρου ευρωπαϊκές εταιρείες. Ήταν λοιπόν ένα από τα λεγόμενα εμπορικά προγράμματα. Η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας όμως ήταν ότι η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια δεν μπορούσε να εφαρμοστεί σε αγωγό αερίου με σημείο εισόδου σε τρίτη χώρα και σημείο εξόδου εντός της Ευρώπης. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή κάνουμε δύο πράγματα. Αφενός πρέπει αμέσως να αλλάξουμε την νομοθεσία μας ώστε όλες οι ρυθμίσεις της αγοράς αερίου να ισχύουν και στο υπεράκτιο κομμάτι, στο κομμάτι που αφορά τρίτες χώρες. Από την άλλη όμως, σε περίπτωση που δημιουργηθεί ο αγωγός Nord Stream, να ταιριάζει στην ε, τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα εγκριθεί από το Συμβούλιο ή όχι, αλλά αυτό που λέει η νομική υπηρεσία είναι ότι δεν μπορεί να βασιστεί σε νομικό κενό. Να έχουμε έναν αγωγό χωρίς ρύθμιση ή που να ρυθμίζεται αποκλειστικά από την ρωσική νομοθεσία και να εισέρχεται στο έδαφος της Ευρώπης. Γνωρίζετε καλά πάντως ποια είναι η γνώμη μου για το Nord Stream 2. Το άλλο που κάνουμε στην αγορά αερίου είναι ότι εξετάζουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για το αέριο. Διότι πρέπει να ρυθμίσουμε τις αγορές, ε, μάλλον έχουμε ρυθμίσει τις αγορές ε, ηλεκτρισμού, δεν έχουμε όμως κάτι αντίστοιχο στο αέριο. Έχουμε λοιπόν ε, εκπονήσει μελέτη που εξετάζει πώς λειτουργεί το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για το αέριο στην Ευρώπη και πώς θα λειτουργήσει στο ε, μέλλον ε, και έχουμε διαβούλευση με ε, διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της μελέτης θα εξετάσουμε αν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των κανόνων για το φυσικό αέριο, διότι δεν συμπεριλαμβανόταν στο πρόγραμμα εργασίας. Προχωρήσαμε πολύ γρήγορα στα υπόλοιπα θέματα και μάλλον και αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να το εξετάσουμε. Όσον αφορά ε, ε, τους σταθμούς φόρτισης, τους κανονικούς ε, και τους υψηλής ταχύτητας. Όσον αφορά το θέμα αυτό, σας παραπέμπω στην οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα και η κανονική σταθμή φόρτισης και η υψηλή ταχύτητας. οι κανονικοί ε, έχουν ισχύ μέχρι 20 κιλοβάτ, ενώ οι υψηλής ταχύτητας έχουν 22 ε, και έχουν, λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα. Μάλλον δεν θα αρκεί η παρούσα υποδομή, αλλά θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Μάλλον κάποιος θα παράσχει τους σταθμούς αυτούς, διότι θα συμφέρει από επιχειρηματική άποψη. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ας ετοιμάσουμε το έδαφος σε περίπτωση που κάποιος θέλει να φορτίσει το αυτοκίνητό του στο σπίτι του. Στα κτίρια που έχουν πάρκινγκ. σε δημόσιους χώρους. Σίγουρα μπορούμε να έχουμε τα δύο είδη σταθμών φόρτισης. Και εάν έχουμε τους κανονικούς σταθμούς σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να φορτίσει κανείς ε, πλήρωσε την ε, μπαταρία, μπορεί να φορτίσει αρκετά ώστε να φτάσει σπίτι του. Αλλά στους αυτοκινητόδρομους Εκεί χρειάζεται υψηλή τάση για να μπορέσει κανείς να φορτίσει πιο γρήγορα. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Αλλά όλοι λέμε ότι θέλουμε ηλεκτροκινητικότητα, κάτι που δεν μπορούμε να πετύχουμε αν δεν έχουμε σταθμούς φόρτισης. Και θα πρέπει να τους δημιουργήσουμε. με λογικό ρυθμό, με ευρωπαϊκή στήριξη, με στήριξη των κρατών μελών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε όμως την υποδομή. Αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο να μειώσουμε τις εκπομπές μας. Απλά με μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, διότι θα είναι αδύνατον για τους κατασκευαστές ε, να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις χωρίς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τέθηκε ερώτηση σχετικά με το ε, σχέδιο που προτείναμε και έχουμε χρησιμοποιήσει μελέτη του Πανεπιστημίου της Αθήνας και η οποία στηρίχθηκε στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία όταν έγινε η προσωμείωση. Και μάλιστα στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις τεχνολογίες ενέργειας. Κάποιοι ευρωβουλευτές έχουν επιστήσει την προσοχή μας στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές στο κόστος της ενέργειας. Γι' αυτό ζητήθηκε να αξιολογήσουμε τα σενάρια με τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές ε, και σε σχέση με τον στόχο ε, ενεργειακής απόδοσης κατά 30% και 33% ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, καθώς ε, και με 33% και 45% αντίστοιχα. Και επίσης ε, στην ερώτησή σας απαντώ ότι προχώρησα όσο μπορούσα εντός του σώματος των επιτρόπων για να πετύχουμε συμβιβασμό. Και μάλιστα πήγα και πιο πέρα από αυτό που ήθελε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενεργειακή απόδοση. Στους τριμερείς διαλόγους θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε ποια είναι η θέση μου. Αλλά, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά να εξετάζουμε και την αναλογία κόστους-όφελους. Να εξετάζουμε και την οικονομική αποδοτικότητα. Δεν ε, θέλουμε να υπονομεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Προσωπικά, δεν έχω πιστεί ότι η καινοτομία θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από τους στόχους που θέτουν οι πολιτικοί. Μπορεί να υπάρξουν ε, ε, επαναστάσεις ε, στην καινοτομία, θα υπάρξουν και μειώσεις του κόστους. Όταν μιλώ για χαμηλές εκπομπές, δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το υδρογόνο οι κυψέλες υδρογόνου αποτελούν επίσης σημαντικό τμήμα του θέματος αυτού. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Τούρμες, προσπαθούμε να πετύχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, να έχουμε νέους ε, κανόνες ε, κατά προτίμηση εντό του Ιουλίου. Έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα αυτό, διότι εάν μπορέσουμε να έχουμε συμβάσει για την ενεργειακή απόδοση, θα πετύχουμε τελείω άλλα επίπεδα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και θα έχουμε τεράστιες δυνατότητες για ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, διότι η ομορφιά των προγραμμάτων ενέργειας είναι ότι είναι μικρά προγράμματα ε, κατάλληλα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργούν πολλές θέσεις απασχόλησης, είναι κάτι λοιπόν που στηρίζουμε. Τι σημαίνει όμως αυτό για την Ισπανία, διότι συνομιλήσατε με την Ισπανική κυβέρνηση. Θα λύσουμε το πρόβλημα της Eurostat, θα έχουμε θετική ανταπόκριση από την Ισπανία. Ένα χρόνο προσπαθήσαμε να το συζητήσουμε. Προσπαθήσαμε να πείσουμε τον κόσμο με τις κατευθυντήριες γραμμές, με τα, τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Προσπαθήσαμε να πείσουμε για τα ωφέλη τους, τα πλεονεκτήματά τους και υπονοούμε και τους νέους κανόνες ε, για τα λογιστικά πρότυπα. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά δίνουμε τη μάχη μας. Τέθηκε και μία άλλη ερώτηση. Είπατε ότι δεν είναι σαφής η διαφορά κοστος ωφέλους για κάποιο από τα μέρη. Αλλά εδώ έχουμε δύο στοιχεία. Το κόστος και το όφελος, αλλά και το θέμα της, ενεργεια... της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και θα πρέπει να εξορροπήσουμε τα δύο στοιχεία. Πάντως δίκιο έχετε, μερικά σχέδια πρέπει να γίνουν αλλά κάνουν δύσκολη τη ζωή και την τρομολόγηση των σχεδίων αυτών κάποιοι διοικητικοί περιορισμοί. Κύριε Ζωχρίνιο, ε, θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για την τραγική απώλεια ζώων και τα πολύ άριθμα θύματα που είχαμε στη γειτονική μας χώρα, την Πορτογαλία, που μαστίζεται τακτικά από πυρκαγιές. Τέτοιου είδους περιστατικά όχι μόνο μας θλίβουν, αλλά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της συνεργασίας και επέμβασης και αλληλοβοήθειας όταν σκύπτουν τέτοιες καταστροφές. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και η διακυβερνητική αλληλεγγύη και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και ξέρουμε πώς η παγκόσμια θέρμαση, ε, η θέρμαση του πλανήτη επηρεάζει και την κατάσταση αυτή. Είπατε ότι έχουμε το θερμότερο καλοκαίρι της δεκαετίας και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου, στις μεσογειακές χώρες, το κύμα του καύσωνα πραγματικά μας πλήττει και υποφέρουμε από αυτό. Και σίγουρα η ενεργειακή διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του πακέτου. Θα έχει νευραλγική σημασία. Γιατί αν υιοθετηθούν οι εθνικοί στόχοι, πάει καλά η διακυβέρνηση και δεν θα κινητοποιηθεί η διαδικασία επί παραβάση. Ε, όταν έχουμε δεσμευτικούς στόχους όμως, βολιδοσκοπούμε τα κράτη-μέλη για το επίπεδο φιλοδοξιών τους και βλέπουμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί ο γενικός στόχος, ο κοινοτικό. Γι' αυτό και η διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική και ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί εθνικά δεσμευτικούς στόχους, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνα το Συμβούλιο. Πάντως σίγουρα η διακυβέρνηση έχει κέριο ρόλο. Φανταστείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει σε σημαντικούς κλάδους όπως οι μεταφορές, η γεωργία και τα κτίρια. Εκεί έχουμε εθνικούς δεσμευτικούς στόχους, οπότε στη διακυβέρνηση θα δούμε ποια είναι η πρόοδος σε επιμέρους τομείς για να υλοποιηθούν αυτοί οι γενικοί εθνικοί στόχοι. Οπότε η ενεργειακή διακυβέρνηση θα έχει θεμελιώδη σημασία. Και στην ε, Κομισιόν είχαμε δύσκολη πορεία στην αρχή είχαμε κάποια στοιχεία διακυβέρνηση. Ε, επιχειρήσαμε να την ενισχύσουμε και ξέρω ότι και εσεί και ο κύριος Τουρμές ε, είστε υπέρ μιας πραγματικά ισχυρή διακυβέρνηση. Και πιστεύω τελικά ότι θα έχουμε μια διακυβέρνηση που θα ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία του Παρισιού. Πάντως ε, η διακυβέρνηση θεσπίστηκε για να ευθυγραμμίσουμε τις πενταετής περιόδους με την τελική συμφωνία και συμμετείχαμε και στον απολογισμό και έχουμε και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική 50 που επίσης ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία του Παρισιού. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι η ενεργειακή διακυβέρνηση θα αποτελέσει θεμελιώδες ε, εργαλείο και θα παρακολουθήσει του κύκλου και τη Συμφωνία του Παρισιού. Και εκεί έχουμε ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό για να τηρήσουμε τι υποσχέσει μα και μάλιστα ε, στην πορεία να ε, αυξήσουμε και τι φιλοδοξίε μα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι αρκετά περίπλοκο, αλλά δεν είναι το μόνο περίπλοκο ζήτημα στη συζήτηση. Πάντω η Μαλτέζικη Προεδρία σε κάποια σημεία μείωσε το επίπεδο φιλοδοξιών στην ενεργειακή απόδοση, ε, για την υποδομή για τη φόρτιση ε, θα εμείνουμε σε αυτό το θέμα, είναι 95% το ότι προτείνουμε και πιστεύω ότι θα τηρήσουμε και τις υποχρεώσεις μας για πολλή έκθεσης στα πλαίσια του, της σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα και θα ευθυγραμμιστούμε και τη Συμφωνία του Παρισιού ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο αναλυτική αλλά και σε βάθος παρουσίασή σας και για τις απαντήσεις σας. Και είμαστε πεπισμένοι ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσε οι συναντήσει μας πάντα. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα τη μέρης διάταξη. Θα παρακαλέσω να με αντικαταστήσει ο κύριο Ρούμπιχ γιατί πρέπει να συμμετάσχω σε μία άλλη εκδήλωση. Γιατί για Ρωμήρα από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να με αντικαταστήσει. Ναι, όχι. Παρακαλώ. Who's the lady of the method? The, was of the method. The lady who was of, of method. Äh, Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον κύριο Επίτροπο που μας ε, επέτρεψε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το 15. Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Αναδιατύπωση. Θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Στις 16 Φεβρουαρίου η κυρία Ντελκαστίγιο μας υπέβαλε ήδη την έκθεση και στις 23 Μαρτίου επίσης ε, το συζητήσαμε είχαμε πάνω από χίλιες τροπολογίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες επίσης οι αλλαγές που προτείνουν η Κούλτ και άλλη μια επιτροπή και να δώσω το λόγο στην κυρία Δελκαστήγιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό το θέμα αυτό για την ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία σε κάθε επίπεδο. για να αξιοποιήσουμε όλες τι δυνατότητε που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Η συνδεσιμότητα είναι πολύ σημαντική. Είχαμε την πρόταση επιτροπή που τονίζει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι υποδομές. Και ότι χρειαζόμαστε έως και 100 δις για να αναπτύξουμε αυτήν την υποδομή και αυτό βεβαίως ε, θα έχει και τις επιπτώσεις του στο ρυθμιστικό πλαίσιο όπου χρειάζεται ανταγωνιστικότητα, συμβατότητα και μακροπρόθεσμες επενδύσεις για να έχουμε μια ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οπότε, να θέσω το πλαίσιο, να το επενθυμίσω και τους κύριους στόχους μας που θέλουμε να επιτύχουμε με αυτόν τον κανονισμό. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν, πρώτα απ' όλα τους Κιώδης. Όλοι με βοήθησαν, με πολύ επικοδομητικό τρόπο, που είναι βεβαίως ε, αναγκαία η συνεργασία για να προωθήσουμε τέτοια θέματα. Οι προτάσει τους ήταν πάντα ευφυεί και ενδιαφέρουσε και στον ένα τον άλλο βαθμό συμφωνώ. Αλλά όλες οι προτάσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά και οι, οι οι συνεργάτες μας από τις ομάδες μας και η γραμματεία της Ήτρε με βοήθησαν πάρα πολύ. Καταπληκτική ήταν. Θέλω να το τονίσω. Και τώρα να περάσω σε μερικά βασικά θέματα. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ως εξής. Η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 11 Ιουλίου. Η ΙΜΚΟ ήταν να ψηφίσει σήμερα, αλλά ζήτησε να αναβληθεί η ψηφοφορία γιατί δεν προλάβαιναν. Οπότε η ΙΜΚΟ θα ψηφίσει στις 4 Σεπτεμβρίου και εμείς θα ψηφίσουμε στις 11 Σεπτεμβρίου. Ε, δεν είναι και μεγάλη καθυστέρηση γιατί ανάμεσα είναι οι θερινές διακοπές. Και την τελική απόφαση τελικά θα ληφθεί ως εξής. Η τελευταία συνάντηση των σκιωδών θα γίνει στις 11 Ιουλίου. Θα υπάρξει άλλη μία την επόμενη εβδομάδα. Τώρα τι πρόοδος έχει σημειωθεί. Μας αφής πρόοδος για το φάσμα, αναμφίβολα. έχουμε έναν προκατακτικό συμβιβασμό, α το πω έτσι, γιατί συμβασμός είναι όταν όλα έχουν αποφασιστεί, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο για όλα τα θέματα που αφορούν το φάσμα, που είναι ο πιο σημαντικός τομέας, μαζί με την πρόσβαση βέβαια. Έχουμε συμφωνία και για τον ορισμό του δικτύου πολύ υψηλής ικανότητας. Έχοντας αυτόν τον ορισμό, πρέπει μετά να τον αξιοποιήσουμε για να είναι συμβατά όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την πρόσβαση. Γιατί μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό ορισμό του VHCN, αλλά αν δεν υπάρχει η σωστή υποδομή για την πρόσβαση για να προσελκύσουμε επενδύσεις και για να υπάρχει προβληψιμότητα και βεβαιότητα, τότε ναι, μεν θα έχουμε καλό ορισμό, αλλά έτσι σκέτο. Έχουμε λοιπόν ε, μία προκατακτική συμφωνία για το φάσμα και τώρα λοιπόν θα ασχοληθούμε κυρίως με την πρόσβαση. Τίθεται μια σειρά από θέματα, το βασικό μοντέλο επενδύσεων, και σε τι βαθμό θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το μέσο που προτείνει η Κομισιόν για να να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί αυτό το VHCAN. Έχουμε επίσης τις ε, συμμετρικές υποχρεώσεις και διάφορα άλλα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα μη ανταγωνιστικά ολιγοπόλια που δεν είναι πρόβλημα τώρα για την Ευρώπη. Ίσως ε, να είναι πρόβλημα σε μία ή μερικές χώρες, αλλά γενικά όχι. Αλλά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα με τους συντονιστές, με τους σκιώδες, συγγνώμη. Και φυσικά θα σημειώσω ό,τι πείτε. Και ό,τι μου πείτε και τώρα βεβαίως ε, θα το λάβω υπόψη μου να δω πώς μπορώ να το εντάξω στη γενική μου προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία πέτρα νάτρια από το S&P για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά αρκούν, διότι ήταν πολύ καλή η εισαγωγή της εισηγήτριας ε, Καστήλιο. Να προσθέσω κάποια πράγματα. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που κινούμαστε τόσο γρήγορα. Το Συμβούλιο κινείται πιο αργά όπως ακούσαμε και επίσης ε, η ΙΜΚΟ ήθελε περισσότερο χρόνο. Θα το εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό και εμείς στην Επιτροπή μας. Πάνω από χίλιες τροπολογίες είχαμε, το οποίο σημαίνει ότι όλοι διάβασαν προσεκτικά την πρόταση και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που στοχεύουμε. Θέλουμε ψηφιακή υποδομή, ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η οικονομία των δεδομένων στην Ευρώπη, η οικονομία των gigabit. Και στο πλαίσιο αυτό δεν κάνουμε απλά τα συνηθισμένα, θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο και να βρούμε τρόπο να αυξήσουμε τις επενδύσεις ε, στα πολύ υψηλή χωρητικότητα σε δίκτυα. Και υπάρχουν κάποια άλλα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για τις επενδύσεις, όπως είναι το φάσμα, τα επιχειρηματικά μοντέλα και η πρόσβαση. οι αγορές αυτές ήδη υπάρχουν. Θέλουμε η ανταγωνιστικότητα να καθοδηγεί τις επενδύσεις ε, και φυσικά και την ζήτηση. Είδαμε ότι έχουμε πάνω από 20 διαφορετικές προτάσεις εδώ στην Ευρώπη γι' αυτό. Ε, θα δούμε τις ε, εξελίξεις αυτές, θα δούμε τα δίχτυα πέμπτης γενεάς. Ε, δεν ανησυχώ όσον αφορά την ζήτηση για τις υποδομές. Ως πολιτική όμως δεν θέλουμε ψηφιακό χάσμα στην Ευρώπη. Θέλουμε αντιθέτως το σύνολο της Ευρώπης να αποτελεί μια ψηφιακή αγορά και ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι σημαντικό πολιτική αυτό να πετύχουμε. Και θα δημιουργηθεί ψηφιακό χάσμα, να σας θυμίσω, αλλά θέλουμε να το αποφύγουμε. Θα πρέπει όλοι να έχουν γρήγορη σύνδεση σε λογική τιμή και αυτό αποτελεί μέρος του πακέτου αυτού. Και αυτό αποτελεί βάση για όλους, όχι μόνο για τους καινοτόμους επενδυτές. Κλείνοντας, η πρόταση αυτή ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται κάποια ρύθμιση ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική η αγορά και να μην έχουμε εκ νέου μονοπόλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευσέντο Σενόφσκι από το ECR, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν. Είναι τεράστιο αυτό το πακέτο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε σημαντική ευθύνη, διότι η αγορά αναπτύσσεται ραγδαία και είναι πολύ δύσκολο να την ποσοτικοποιήσουμε οικονομικά. Γι' αυτό χαίρομαι πολύ με την ανοιχτή συζήτηση που έχουμε και εκτιμώ ιδιαίτερα τα όσα έχει πετύχει η συνάδελφος. Η κυρία ε, Πιλάρ Τελκαστήλιο έχει λάβει υπόψη της ε, όλες τις πτυχές και ο μεγάλος αριθμός τροπολογιών δείχνει πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα αυτό. Επίσης, εκτιμώ το πώς η κυρία ε, Τελκαστήγιο ασχολείται με τα δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και το θέμα της πρόσβασης. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα. Στα περισσότερα θέματα μπορώ να συμφωνήσω με την εισηγήτρια και χαίρομαι που βλέπουμε να υπάρχουν λύσεις για το μέλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως διαφέρουν οι θέσεις μας. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις ε, δυνατότητες προσφυγής για, τους, για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, όπως και για το φάσμα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για 28 διαφορετικές αγορές και υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Πιστεύω όμως ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση. Και η τελική μου παρατήρηση έχει να κάνει με την επικάλυψη με το θέμα του ΠΕΡΕΚ, του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο, διότι καταφέρνει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στα δύο αυτά θέματα. Πρέπει να προχωρήσουν τα δύο θέματα αυτά μαζί δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο και πρέπει να συνάδουν μεταξύ τους. Γι' αυτό προσπαθούμε επίσης να συντονίσουμε τα χρονοδιαγράμματα και γι' αυτό ελπίζουμε στις 11 Σεπτεμβρίου να εγκριθούν και οι δύο αυτές εκθέσεις μαζί. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για τη συνεργασία σας κύριε Καστίγιο και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε πολύ καλή πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Εύσεν. Κάλια Κάλλας από την Άλτε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια, την κυρία Δελκαστήγιο, για την προσπάθειά της. Είναι όντως ευρύτατο θέμα και πλειάδα οι τροπολογίες. Εγώ θα επικεντρωθώ στις συμβαστικές τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά το φάσμα, δεν υπάρχει με ιδιαίτερη διάσταση απόψε. Συμφωνούμε ότι θέλουμε ενοποιημένη πολιτική για το φάσμα, αλλά και κάποιο βαθμό βεβαιότητας για τους ε, κατόχους αδειών φάσματος. Και η διάρκεια τουλάχιστον 25 χρόνων θα πρέπει να αναφέρεται στην ενδιάμεση αξιολόγηση για να μεγιστοποιηθεί η χρήση του φάσματος ε, υπό το φως και της τεχνολογικής εξέλιξης. Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο πρόσβασης, και αυτό είναι σημαντικό, στις συμβαστικές λύσεις δεν ε, είχαμε αρκετά θεαματική πρόοδο. Είπα, καλό θα ήταν να έχουμε ξεχωριστό τίτλο για τα δίκτυα πολύ μεγάλης χωρητικότητας, γιατί ε, Πολλέ χώρες έχουν ε, στόχο μέχρι το 2025 να έχουν πλήρη ανάπτυξη των δικτύων πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Οπότε ίσως ε, καλό θα ήταν να έχουμε διαφορετικές διατάξεις. Επίσης δεν πιστεύω ότι για το λιανεμπόριο η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι φορά την ανάλυση των αγορών είναι σωστή. Καλό θα ήταν να μην έχουμε ε, νομική απέτηση για κάτι τέτοιο σε επίπεδο λιανεμπορίου για την ανάλυση της αγοράς. Ε, σε ό,τι αφορά τις αγορές χοντρικής. Για τα ολιγοπόλια να αντιμετωπίσουμε αυτή την τάση, αλλά αν η κυρία Δελκαστήγιο ε, επιμείνει στη θέση της, ε, να μην υπάρχει ρύθμιση για τις επενδύσεις, ίσως έτσι αυξηθεί ο κίνδυνος των λιγοπολίων. Δεν είμαι λοιπόν υπέρ της ρυθμιστικής ανάπαυλας για τα μοντέλα ολικών επενδύσεων και ταυτόχρονα να μην έχουμε τίποτα για τα ολιγοπόλια. Ε, μια και η είναι αρμόδια για τους ορισμούς, παρόλο που είναι κατά της αναθεώρησης τους η κυρία Πιλάρ Καστίγιο. πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δεν θεωρώ ότι η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτυχε στο στόχο τη εμβάθυνση τη ενιαία αγορά για τι τηλεπικοινωνίε. Γι' αυτό το θέμα τη ενιαία άδεια για του ε, διασυνοριακού παρόχου θα πρέπει να το εξετάσουμε. Θα ήταν κρίμα να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και να μην ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Γι' αυτό και θα καταθέσω σχετικές συμβαστικέ τροπολογίες αυτά και προσβλέπω σε συνεργασία και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ράιμον δεν είναι εδώ. Η FTD. Ντάβιτ Μπορέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες με στόχο την ε, πρόθεση του ανταγωνισμού και στις υποδομές αλλά και στην παροχή υπηρεσιών. Για την υλοποίηση της ε, ψηφιακής ενίας αγοράς θα πρέπει να έχουμε κατά νου τα συμφέροντα των πολιτών. Αυτό θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης και φυσικά και θεμητό ανταγωνισμό. Μόνο με θεμητό ανταγωνισμό θα γίνουν επενδύσει. 40% μόνο των ε, κατοίκων της υπαίθρου έχουν πρόσβαση στο δίκαιο. Κάτι που είναι θεμελιώδης δικαίωμα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ευρυζωνικότητα παντού, ακόμη και στις ε, πιο φτωχές οικογένειες και στον αγροτικό πληθυσμό. Κάποιες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβάλλουν στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές επιπλέον υποχρεώσεις. Αυτό απαιτεί ο φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όμω έτσι θα στερηθούν κάποιε αρμοδιότητε για να καταπολεμήσουν μονοπόλια και ολιγοπόλια. Θέλουμε να προβλέψουμε τα εχέγγυα ώστε οι εθνικέ αρχέ να μπορούν να συνεχίζουν να προωθούν την ανταγωνιστικότητα προ όφελο των και θα πρέπει οι ρυθμιστικές αρχές να έχουν ένα ε, ευρύ οπλοστάσιο ε, για να καταπολεμήσουν αθέμητες πρακτικές. Επίσης, ε, θα πρέπει να επιτρέπεται ηλική πρόσβαση. Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι το πρώτο μέσο που θα επιτρέπει διαρκή θεμητό ανταγωνισμό και επενδύσεις ε, στις ε, υπηρεσίες αυτές. Για το φάσμα, καλό θα ήταν να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να έχουμε καλύτερη διαχείριση και συντονισμό στο φάσμα. Έχουμε τις ενδιάμεσες βέβαια άδειε, αλλά ξέρουμε τι θα κάνει το Συμβούλιο στον τριμερή διάλογο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο φιλόδοξοι εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως τις μη κερδοσκοπικέ οργανώσεις που κινδυνεύουν να αποκλειστούν. Θα πρέπει οι εθνικές αρχές, ή μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υιοθετήσει πιο φιλόδοξη στάση στην ψηφοφορία τη 11 η Σεπτεμβρίου γιατί μόνο με ένα τέτοιο ευρωπαϊκό κώδικα θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε τηλεπικοινωνίε ε, που θα στηρίζονται σε βιώσιμο θεμητό ανταγωνισμό, θα προστατεύουν τι επενδύσει και ταυτόχρονα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει και μια ανάλυση αντικτύπου στον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις επενδύσεις των παρόχων, να μην αφήσουμε να εκμετάλλευτε αυτή την ευκαιρία και να επιτρέψουμε σε όλου του ε, πολίτες πρόσβαση σε συνδεσιμότητα χωρί όρια με βάση υποδομές και ευρυζωνικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο τον λόγο. Να ρωτήσουμε λοιπόν τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Βέζα Τιαράμπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ την Επιτροπή σας για την πρόοδο που σημειώθηκε για το θέμα αυτό. Που είναι τόσο ευρύ. Ιδιαίτερα για το πλαίσιο. Χαιρόμεθα. Για τη σύγκληση απόψεων που έχει σημειωθεί από ό,τι βλέπουμε στα πλαίσια της Επιτροπής σας και η οποία σύγκληση συγκλίνει και με τις απόψεις της ε, Επιτροπής. Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι τροπολογίε από ό,τι βλέπουμε βοηθούν να διευκρινιστεί το κείμενο που υποβάλαμε και ενισχύουν μερικές βασικές αρχές. <coughs> Συγκεκριμένα. Αυτό που ανέφερε η κυρία Κάλλας για τις άδειες, για την ε, δημιουργία αδειών. Χαιρόμεθα που το Κοινοβούλιο συμμερίζεται τη φιλοδοξία της Επιτροπής να χορηγηθεί νομική βεβαιότητα για τις επενδύσεις στα ασύρματα δίκτυα. Αυτό είναι όλο και πιο σημαντικό όταν ε, αναπτύσσαμε τα προηγούμενα δίκτυα, γιατί τα δίκτυα 5G είναι πολύ πυκνά και χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις για την μεσοπρόθεσμη, για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Όσο περισσότερη, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της άδεια, τόσο σημαντικότερο είναι να έχουν τις δυνατότητες να επέμβουν οι αρχές αν κάτι πάει στραβά. Θεωρούμε ότι η πρότασή μας ήδη περιέλαβε ένα μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Φυσικά μπορεί να ενισχυθεί αυτός ο μηχανισμός. Συμφωνώ πλήρως. αλλά ίσως ε, δεν είναι πιο κατάλληλη η στιγμή για μια τέτοια ενίσχυση ή ενδιάμεση αναθεώρηση. Οι άδειε τώρα χορηγούνται για 15 με 20 χρόνια κατά μέσο όρο και ο υπάρχον μηχανισμός δεν έχει εμποδίσει τις αρχές να διαχειρίζονται πολύ καλά το σύστημα. Αυτό ήθελα να σημειώσω. Τώρα για την πρόσβαση. Φυσικά χαιρετίζουμε και εδώ την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Από ό,τι καταλάβαμε, οι συζητήσεις ε, για τα δίκτυα ολύψηλης δυνατότητας ε, δυναμικού έχουν προχωρήσει και πρέπει να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι για τον ορισμό αυτό. Ο ορισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες συνδεσιμότητας που θα προκύψουν στο εγγύς μέλλον. Αυτό ήταν το σημείο αφετηρίας και για την Κομισιόν για την πρόταση που έκανε για τον ορισμό και από ό,τι καταλαβαίνουμε συμμερίζεστε την άποψή μας. Και φυσικά τα δίκτυα αυτά. Δεν θα είναι μόνο με σταθερές εγκαταστάσεις για το 5G και τα σύρματα δίκτυα θα είναι πολύ σημαντικά. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην απόφαση. Για τη ρύθμιση των αγορών τώρα και ε, επαρκείς εγγύησεις για τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις. Σταθερή μας πεποίθηση είναι ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Η πρότασή μας λοιπόν βασίζεται στο υπάρχον ε, πλαίσιο S&P που έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει, ότι είναι ευέλικτο και μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα στη λειτουργία των αγορών, θέματα ανταγωνισμού. Αλλά δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε. Πρέπει να έχουμε και τα εργαλεία στα χέρια μας για να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο καθυστέρησης ε, της εγκατάστασης αυτών των δικτύων υψηλής, υψηλού δυναμικού. Ιδιαίτερα στις περιοχές που αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες δυσχέρειες για να αποφευθεί αυτό που είπε η κυρία Κόμπουλα Νάτρη, να μην υπάρξουν ψηφιακά χάσματα. Γι' αυτό υπάρχουν κίνητρα στην πρότασή μας για να, γι, να εγκατασταθούν αυτές οι υποδομές. Πρέπει να μείνουν λοιπόν αυτά τα κίνητρα. Πρώτα απ' όλα βέβαια ο κανονισμός πρέπει να βασίζεται σε μια σωστή ανάλυση της κατάστασης των αγορών. Σε κάποιες ε, ιδιαίτερες περιοχές το βασικό είναι οι χρήστες να έχουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Αλλά να τονίσω κάτι άλλο, γιατί ίσως να έχει υπάρξει κάποια παρανόηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, οι ρυθμιστικές αρχές να εξετάζουν τις αγορές λιανικής και να κάνουν αναλύσεις S&P. Δεν είναι στην πρότασή μας. Και κάτι άλλο σημαντικό. Οι κανόνες για τα συμμετρικά αντίμετρα. για τις μετρικές υποχρεώσεις καλύτερα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν, αλλά πρέπει να έχουν και όρια. Θέλουμε να δώσουμε επαρκή κίνητρα στους νέους επενδυτές ε, που θα δημιουργήσουν τα νέα δίκτυα οπτικών ινών. Αυτά είναι τα κύρια σημεία. Να σας ευχαριστήσω για την πρόοδο που έχει σημειωθεί, για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα από το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο και εμείς ως Επιτροπή είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Πρόεδρος. Η Πιλάρα θέλει να πει τίποτα. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προθυμία της και τη διάθεσή της να μας βοηθήσει στην εξέβρεση τεχνικών λύσεων σε κάποιους από τους προβληματισμούς μας. Υπάρχει καλή βούληση και γι' αυτό την ευχαριστώ. Και όπως είπα ήδη στην αρχή, Σημειώνω όλα όσα επεσήμαναν οι συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και είμαι πεπισμένη ότι θα ανταποκριθούμε στο επίπεδο των προσδιοκών και ότι θα λάβουμε τις σωστές αποφάσεις ώστε να πετύχουμε την διασυνδεσιμότητα που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να έχει παγκόσμια διάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πιλάρ. Θα ήθελα να πω ότι θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία στην Ήτρε στις 11 Σεπτεμβρίου. Η ΙΜΚΟ έτσι έχει ακόμα χρόνο να υποβάλει τη γνωμοδότησή της. Προχωράμε στο επόμενο θέμα, που είναι ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η συγητής είναι ο Εύσεν Τοσενόφσκι. 441 τροπολογίες έχουμε και συμβιβαστικές τροπολογίες θα υποβληθούν που θα καλύπτουν όλες τις πτυχές του θέματος αυτού. Δίνω λοιπόν κατευθείαν τον λόγο στον Εύσεν για 5 λεπτά για να μας εξηγήσει τη θέση του. Παρακαλώ Εύσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέρφους μου, τους σκιώδεις εισηγητές, για τη συνεργασία μας. Οι αρχικές μας θέσεις ήταν πολύ διαφορετικές. Είχαμε αρκετές συναντήσεις και εκτιμώ τον ε, ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων που είχαμε. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου, ε, μαζί δηλαδή με την πρόταση για τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Και όπως υπόθηκε, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ε, σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές προτάσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία θα, θα βασιστεί η συμβαστική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των ε, εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Θα πρέπει να είναι πιο καλός ο συντονισμός σε όλη την Ευρώπη. Από την άλλη μεριά είχαμε πολύ καλές εμπειρίες ε, από την ε, παρούσα λειτουργία του ΠΕΡΕΚ, του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Και στο Κοινοβούλιο ε, έχει πολύ καλή φήμη ο φορέας αυτός για την επιρροχνωμοσύνη του. και για την θέση που έχει λάβει σε θέματα που σχετίζονταν με την διαμόρφωση της νομοθεσίας. Το βασικό θέμα που έχουμε μπροστά μας είναι εάν θα πρέπει να συγχωνεύσουμε το ΜΠΕΡΕΚ με την υπηρεσία ΜΠΕΡΕΚ που είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αν θέλουμε να διατηρήσουμε την παρούσα διτή θεσμική δομή η οποία πιστεύω ότι ήταν επιτυχής μέχρι τώρα και που όπως είπα έχει αποκτήσει πολύ καλή φήμη. Ως εισηγητής ε, χαίρομαι που καταφέραμε να πετύχουμε πλειοψηφία υπέρ μια πιο συντηρητική προσέγγισης, να διατηρήσουμε δηλαδή κάποια τμήματα της διτής αυτής δομής. και να την ενισχύσουμε με βάση τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει και την κατάσταση των πραγμάτων. Όσον αφορά τον ίδιο τον Μπέρεκ θα αναβαθμιστεί. θα λάβει νομικό πρόσωπο και έτσι σεβόμαστε τη θέση του Κοινοβουλίου που αποτελεί αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τον κώδικα. Ενώ ο Μπέρεκ θα λάβει νέα αρμοδιότητα και θα μπορεί να λαμβάνει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις. Αυτό λοιπόν έχει συμπεριληφθεί στην πρότασή μας. Υπάρχει ακόμα το θέμα εάν θα πρέπει να υπάρχει σώμα προσφυγών στον ΠΕΡΕΚ. Το θέμα αυτό εκκρεμεί ακόμα. Πιστεύω όμως ότι θα λυθεί στη σημερινή συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. στην συμβιβαστική μας πρόταση. Έχουμε κάνει πιο αποτελεσματικούς τους κανόνες λειτουργίας ε, του ε, σώματος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου. Και το γεγονός ότι ο Μπέρεκ ε, είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζεται στον νέο τίτλο του Μπέρεκ που είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, για τις ε, Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές ενώ θα διατηρήσουμε και την πιο σύντομη ονομασία ε, το γραφείο Μπέρεκ. Ε, πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα αυτά, κάτι που προσπάθησε να περιορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ΠΕΡΕΚ θα πρέπει να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα, τα οποία απορρέουν από τον κώδικα για την περιαγωγή. Είμαστε διατεθειμένοι να συμπεριλάβουμε το θέμα αυτό στο κείμενο και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη συνάφεια με άλλες, νομοθετικές, με άλλες νομοθεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην χρειάζεται συνεχής τροποποίηση αυτού του κανονισμού. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλά νέα καθήκοντα για τον ΠΕΡΕΚ, ότι αλλάζει η αγορά Πιστεύουμε όμως ότι ο Μπέρεκ θα κάνει καλά τη δουλειά του και επίσης θα ενισχύσουμε τη ρήτρα αναθεώρησης. Μετά από πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει εάν λειτουργεί καλά η διητή δομή ή αν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Νέα καθήκοντα για τον Μπέρεκ σημαίνει επίσης ε, υψηλότερες απαιτήσει από το γραφείο Μπέρεκ και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε και το προσωπικό ε, ώστε να έχουμε 40 ή 45 υπαλλήλους. Πιστεύω επίσης ότι η Μαρία Κάπριελ, η επίτροπος που έχει οριστεί τώρα, έχει μιλήσει πολύ θετικά για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία και προσβλέπω στην συζήτηση με τους κοιόδης εισηγητές στο μέλλον. Και πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε γρήγορα την εξέταση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ευσεν. Επόμενος ομιλητής ε, κανονικά ήταν ο κύριος Κάρινς από το ΕΕΛ και ε, ζητεί συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρόν. Ε, γι' αυτό θα διαβάσω σύντομα τα όσα έγραψε. Ευχαριστώ καταρχήν τον εισηγητή τον κύριο Τσανόφσκι και τους και οδησηγητές για την εξαιρετική προσπάθεια και συνεργασία για την έκθεση. Το θέμα δεν είναι η μορφή του Μπερέκα, αλλά οι του. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις ε, ανάγκες ε, που εξυπηρετεί ο Μπερέκ. Και αυτό να το έχουμε υπόψη στη συζήτηση για τη μορφή που θα λάβει. Και θα πρέπει οι στόχοι του Μπερέκ ε, να πραγματοποιηθούν. Φοβάμαι ότι μια νέα δομή θα αυξήσει τη γραφειοκρατία. Θα πρέπει να δούμε πώς οι φυστάμενες και εύρυθμες δεδομές μπορούν να λειτουργήσουν. Ένα νέος οργανισμό ηλεκτρονικών ε, ε, επικοινωνιών δεν θα είναι πανάκια για να διορθώσουμε τον κατακαιρματισμό στην αγορά. Ε, θέλουμε να στηρίξουμε τις λειτουργίες στο νέο κανονισμό για τον ΠΕΡΕΚ και γι' αυτό θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι νέες ευθύνε και αρμοδιότητες να συμπεριλαμβάνονται και τις διατάξεις για τον προπολογισμό και το προσωπικό της υπηρεσίας του Μπερέκ. Ήδη έχουμε καταλήξει γενική συμφωνία για τα βασικά ζητήματα και η συμφωνία αυτή φαίνεται να είναι ισορροπημένη για τη σχέση μεταξύ του νέου οργανισμού και της υπηρεσίας του Μπερέκ. Θέλουμε, ε, χάρη σε αυτή την ισορροπία, ε, να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτού του, αυτής της πρότασης. Αυτά μας λέει ο κύριος Κάρης και τώρα περάμε στην κυρία Κρέλα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Στην αρχή είχαμε δυσχέρειες γιατί υπήρχε μεγάλη απόκληση των θέσεων. Εγώ είχα την άποψη και η πρότασή μου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει μια καλή πρόταση. Αυτή η κατάρριξη της διπλής δομής να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική και πλήρως ανεπτυγμένη δομή. Αυτός ο φορέας μετά από πολλές συζητήσεις με τον Μπέρεκ, με εθνικές ρυθμιστικές αρχές, με τους Κιώδης, πρέπει να διαπιστώσω όμως ότι δεν έχουμε πλειοψηφία. Χρειάστηκε να διαπιστώσω ότι δεν υπήρχε πλειοψηφία για τέτοια άποψη στο σώμα μας, οπότε πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα υπάρχοντα όργανα για να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Και νομίζω ότι όπως το είπε και ο εισηγητής, αυτό που και εγώ θεωρώ λοιπόν απολύτως αναγκαίο, είναι ναι μεν ναι, να διατηρηθεί η διπλή δομή του Μπέρεκ, αλλά να γίνει ένα νομικό πρόσωπο και να μπορεί να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις. Αυτό θα βοηθήσει είναι ένα σημαντικό βήμα για την ε, εσωτερική αγορά στις ε, τηλεπικοινωνίες και θα αποφασίσουμε τέτοιες τροπολογίες συμβαστικές. Επίσης, πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνέχεια στην εργασία. Οπότε η Προεδρία να παραταθεί στα δύο χρόνια, αυτό βοηθάει η θητεία των Προέδρων. Κάπως έτσι εργάζονται και διάφοροι άλλοι φορείς της Ένωσης Χαίρομαι πολύ που ο Μπέρεκ στο μέλλον δεν θα ασχολείται μόνο με διοικητικά θέματα, αλλά και με θέματα ουσίες. Και θα μπορεί να βοηθά λοιπόν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, μικρότερες χώρες. Συγγνώμη. Και ελπίζω ότι θα έχει και μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ιδιαίτερα το γραφείο του Μπέρεκ, το Μπέρεκ Office, για να έχει και περισσότερους ε, υπαλλήλους και ε, ελπίζω και για αυτό το θέμα να ε, υπάρξει πλειοψηφία μετά από την διατύπωση κατάλληλων συμβασμών από τους ε, σκιώδες. Ευχαριστώ πολύ. άντε τώρα. Η κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Χαίρομαι που δεχτήκατε μερικές από τις τροπολογίες μας, η ανάγκη ο Μπέρεκ να συνεργάζεται με τις αρχές προστασίας των καταναλωτών, και να συμμετέχει στι πρωτοβουλίε για τα ανοιχτά δεδομένα και να είναι το ενιαίο σημείο για ανταλλαγή προφοριών και επαφή μεταξύ των διαφόρων ρυθμιστικών αρχών. Χαίρομαι επίση που ο Μπέρεκ θα έχει θα γίνει νομικό πρόσωπο. Βεβαίως, εφόσον θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες πρέπει να έχει και τις σωστές διαδικασίες. Όμω λυπάμαι που οι συζητήσει για το θέμα αυτό εστίασαν κατά λάθο σε αυτό το φόβο μήπως δημιουργήσουμε, μία τερατώδη αρχή. Φυσικά δεν θέλουμε την γραφειοκρατία και την ε, αναποτελεσματικότητα. Και αυτό κατά τη γνώμη είναι αυτό που υπάρχει τώρα με αυτή τη διπλή δομή μεταξύ του BEREC και του BEREC Office. Αυτό δεν το βλέπουμε σε κανέναν άλλο παρόμοιο φορέα γιατί είναι μη αποτελεσματικό και οδηγεί σε ε, επικάλυψη. Αν υπάρχει νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα, μπορεί να πούμε ότι είναι αρχή, μπορεί να πούμε ότι είναι σώμα, μπορεί να είναι φορέας. Αλλά είναι φορέας της Ένωσης, εφόσον θα, έχει εφόσον θα είναι νομικό πρόσωπο. Τώρα αντί να δώσουμε ε, οντότητα νομικού προσώπου σε ένα φορέα, δίνουμε σε δύο. Γιατί θέλουμε δύο. Ένας φορέας με ένα νομικό πρόσωπο θα ήταν η καλύτερη λύση. Αλλά συμβασμοί αυτό είναι συμβασμοί. Το οποίο σημαίνει ότι δεν συμφωνούν όλοι απόλυτα με αυτούς. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να ολοκληρώσουμε σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η σκιώδη συγκητές. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρία λεπτά. Όλοι μαζί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση για το θέμα αυτό και γνωρίζουμε πόσο ε, δυσκολίες δημιούργησε σε μερικούς για να συμφωνήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά αντιλαμβάνομαι και το λόγο για τον οποίο καταλήξατε στις συγκεκριμένες συμβαστικές τροπολογίες. Λίγα σχόλια μόνο. Χαίρομαι που συμφωνείτε με την απόδοση νομικής προσωπικότητας στον φορέα Μπερέκ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όταν ο φορέας έχει περισσότερες αρμοδιότητες και κυρίως μπορεί να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις, είναι σκόπιμο να έχει και νομική προσωπικότητα. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του από τη στιγμή που αναλαμβάνει και νέε αρμοδιότητε. Σε αυτό συμφωνούμε. Ταυτόχρονα, υπάρχουν κάποια πράγματα που μα θλίβουν. Λυπούμαστε, για παράδειγμα, που καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι η διπλή δομή είναι προτιμότερη από μια ενιαία δομή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια διπλή δομή δημιουργεί περιττή γραφειοκρατία και δεν επιφέρει την αποτελεσματικότητα που θα χρειαστεί στο μέλλον ο φορέας Μπερέκ για να ανταπεξέλθει στις επιπλέον του αρμοδιότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Μπερέκ Office, την υπηρεσία του Μπερέκ, Φυσικά ευθυγραμμιζόμαστε με την ενιαία προσέγγιση, αλλά πραγματικά θεωρούμε ότι είναι κρίμα που το προσωπικό της υπηρεσίας του Μπέρεκ, του BEREC Office, ε, ε, έχει περιορισμένο ρόλο στα τρέχοντα καθήκοντα, δηλαδή να παρέχει υποστήριξη διοικητική στις δραστηριότητες του φορέα Μπερέκ. Είναι με σημαντικό, αλλά θα ήταν προτιμότερο να έχει και ο Μπέρεκ υπηρεσία ένα προσωπικό που θα μπορούσε να επισέρχεται και στο ουσιαστικό έργο και όχι μόνο στο τεχνικό της υποστήριξης. Γιατί στο μέλλον θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες, είπα ο Μπερέκ. Αν δούμε πώς λειτουργεί τώρα ο φορέας, διαπιστώνουμε ότι ανταπεξέρχεται τέλεια. Αλλά οι μικρές ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόβλημα και ζορίζονται για να συμμετέχουν στο έργο. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων που είναι οι ομάδες εργασίας που πραγματικά κάνουν το βασικό ουσιαστικό έργο, βλέπουμε ότι σε αυτές τις ομάδες εργασίας κυριαρχούν λίγες ε, ρυθμιστικές αρχές. Αυτή τη στιγμή 17 ρυθμιστικές αρχές δεν προεδρεύουν σε καμία ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων του φορέα Μπερέκ. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό αν είχαμε έναν οργανισμό με ενιαία δομή, γιατί έτσι θα παρήχαμε στήριξη και στο τρέχον έργο του Μπερέκ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών διεξάγεται συζήτηση για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τον ΜΠΕΡΕΚ ε, και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Επικοινωνιών, την ΕΝΙΣΑ ε, και το, ε, την ΙΣΑ τον τρίτο οργανισμό, ώστε να υπάρχει ένας εξορθολογισμός του έργου και των τριών οργανισμών, που έχουν μεγάλη σημασία στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Ο εισηγητής μας και πάλι, ο κ. Στοσανόφσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους ε, και τους σκιώδης εισηγητές ιδιαίτερος και εκτιμώ ιδιαίτερω ε, την προσέγγιση σας στο θέμα αυτό. Ε, πραγματικά δεν ήταν καθόλου εύκολο να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις και εκτιμώ ιδιαίτερος ε, ε, το σχόλιο της κυρίας Κρέλ για την αναζήτηση της πιο λογικής και ισορροπημένης λύσης. Προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε διστάμενες απόψεις. Εγώ δεν μπόρεσα ε, να συμφωνήσω με τη γνώμη και δεν συμφωνώ ακόμη με, την, με το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η διατήρηση της διπλής δομής θα αυξήσει τη γραφειοκρατία. Διαφωνούμε γιατί ούτως ή άλλως έτσι λειτουργούσε μέχρι τώρα ο φορέας Μπερέκ. Και δεν θεωρώ ότι κάτι που στηρίζεται στην εμπειρία μας ε, και έχει αποδείξει τη σωστή λειτουργία του ε, και χρησιμοποιεί την επαγγελματική γνώση και την περιγνωσία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, μπορεί να ανατραπεί με μια πρόταση για μια ενιαία δομή. Αντιλαμβάνομαι βέβαια τον προβληματισμό και τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και προβλέψαμε ένα μηχανισμό αξιολόγησης και αναθεώρησης μετά την πενταετία για να εξετάσουμε κατά πόσο λειτουργεί εύρυθμα αυτή η πρόταση. Θα έχουμε στο μεταξύ και την ανάπτυξη του κώδικα, γιατί πρόκειται για μια τεράστια αγορά που εξελίσσεται δυναμικά και ραγδαία και είναι αδύνατο να προβλέψουμε από τώρα το μέλλον. Γι' αυτό και προβλέψαμε τη ε, ρήτρα αυτή ε, για την αναθεώρηση. Σας ευχαριστώ θερμά που επιτέλους θα διεκπαιρεώσουμε και αυτό το θέμα, γιατί σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, έχουν μείνει κάποια δευτερεύοντα ζητήματα μόνο εκκρεμή, αλλά ευελπιστώ ότι θα τα διαθετήσουμε και αυτά και θα καταλήξουμε σε κοινή λύση. Όπως είπατε, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα στην αρχή και αυτό και εκτιμώ ιδιαίτερω ε, την συνδρομή των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά πήγε αυτή η συζήτηση, όπως ξέρετε. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Άρα έχουμε ακόμη χρόνο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και μάλιστα νωρίτερα τη συνεδρίασή μας και θα τα ξαναπούμε στις 3 με τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμες. Λοιπόν, καλή όρεξη. Χαίρετε, λήξεις.